Merci. Äh, Δεν ξέρω τώρα με τι σειρά θα αρχίσουμε. Έχουμε ενδιαφέροντες επισκέπτες. Ο προεδρευτής Χέργα Νοβάπνη, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, πίσω να τελειώσω σωστά, ο κύριος Ιβμένη, πρόεδρος του Ερευνητικού Συμβουλίου και ο κύριος Μέκε που έχει επίσης πραγματικά να μας πει για το ε, εκτελεστικό, την εκτελεστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα. Ελπίζω να απαραίτητα σωστά το τίτλο σας. Σας χαιρετίζω όλους εγκαρδιότητα. Τώρα δεν ξέρω με τι σειρά θέλετε να μιλήσετε. Η κυρία καθηγήτρια θα αρχίσει. Πολύ ωραία είναι και νεοεκλεγμένη πρόεδρος και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η καθηγήτρια κυρία Νοβότμη είναι παρούσα. Και τους άλλους χαιρόμαστε επίσης βέβαια. Αλλά έτσι έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε το τι γίνεται στο ε, ε, ε. Έχετε το λόγο κύριε Νοβότμη. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα και μια μεγάλη τιμή να είμαι ενώπιον τη Επιτροπή Βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τελευταία φορά που ήμουν ενώπιον σα ήταν πριν από την έναρξη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα. Έκτοτε έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και χαίρομαι πάρα πολύ που μα προσκαλείτε για αυτή την παρουσίαση. Εν συντομία, θα κάνω μια αναδρομή της ε, ιστορίας των πραγμάτων πριν από την ίδρυση του ΕΣΣ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΕΣΕ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα μάλλον, και θα ήθελα να ανταλλάξουμε απόψει για το πώ θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε καλύτερα αυτό το Συμβούλιο και να το κάνουμε πραγματικά ένα πρώτη τάξεω χρηματοδοτικό ίδρυμα για την έρευνα. Μέχρι στιγμή το Συμβούλιο Έρευνα ήταν μια ιστορία επιτυχιών, όχι μόνο φέτο, αλλά και στο παρελθόν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την επιστημονική κοινότητα και μεταξύ φορέων όπως η ΕΜΑ και σε άλλους χώρους εξάλλου. Το παράδειγμα, όπως θέλουμε να το λέμε, του Ευρωπαϊκού το υπόδειγμα, αν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα έχει την εξή μορφή. Είναι η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνει η χώρα ένα διαγωνισμό για να υποστηρίξουμε τους καλύτερου μεμονωμένου ερευνητέ σε έρευνα εχμής. Μέχρι τώρα αυτή η έρευνα γινόταν, επιβραβευόταν μονάχα σε εθνικό επίπεδο και τώρα αυτό είναι ένα νέο επίπεδο επιβράβευσης. Έχουμε μια πρώτη ε, εξασφάλιση, μια πρώτη μορφή χρηματοδότησης, ένα πρώτο επίπεδο χρηματοδότησης που βοηθάει να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των ερευνητών. Γιατί ένας από τους λόγους απώλειας πολλών ερευνητών είναι ακριβώς αυτός, ότι οι ερευνητές πηγαίνουν στι ΗΠΑ και δεν ξαναγυρίζουν γιατί θεωρούν ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι πράγματι ανεξάρτητοι. Θέλουμε να τους κρατήσουμε αυτούς τους καλύτερους, θέλουμε να επαναπατρίσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει και θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα ελκυστικό χώρο εργασίας και έρευνες. Η έρευνα εχμής σημαίνει και έρευνα στα όρια της γνώσης, ανάπτυξη τεχνολογιών που βρίσκονται στα όρια του επιστητού και πιστεύουμε ότι κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα οδηγήσουν και σε νέες καινοτομίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνα είναι μια ιστορία επιτυχίας γιατί μπορούμε να δούμε ότι είχαμε κάποιο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την επίτευξη νέων προτύπων αξιολόγησης. Να σας δώσω μονάχα ένα παράδειγμα. Για το τελευταίο τέφος του Science αναφέρεται η αναδιάρθρωση του πολωνικού συστήματος αξιολόγησης που θα ακολουθήσει ακριβώς το σχήμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνες. Και πράγματι πάρα πολλοί έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά μας και τα πρότυπά μας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μεταλαπαδευτούν σε όλη την Ευρώπη. Επίσης για πρώτη φορά έγινε πραγματικά ένας διαγωνισμός στον οποίο μια άμυλα μεταξύ πανεπιστημίων η Πριτάνης, ήδη αρχίζουν να αμιλώνται για τον αριθμό χορηγήσεων που έχουν πάρει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Και αυτό προωθεί και τον συναγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων, τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων. Έχουμε ήδη ξεπεράσει ήδη το επίπεδο των χιλίων χορηγήσεων από το Συμβούλιο Έρευνα. Υπάρχει ένα αυξανόμενο αριθμό νέων ερευνητών, πεπειραμένων ερευνητών επίση στην Ευρώπη, που ξεκινούν να σχηματίζουν ένα πραγματικά μοναδικό ευρωπαϊκό ερευνητικό ιστό σε ό,τι αφορά την έρευνα στα όρια της γνώσης. <clears throat> Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στον τομέα αυτό που αφορά τα όρια της γνώσης. Έχουμε επίσης μεταλαμπάδευση γνώσεων που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από άλλους ερευνητές και επίσης έχουμε καταγάγει επιτυχίες στο ότι πολλές χώρες έχουν αναλάβει να χρηματοδοτήσουν και αυτές νέους ερευνητές, τους οποίους εμείς δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε, αλλά που θεωρήσαμε ότι πράγματι ήταν υψηλού επίπεδου, φτάσαμε δηλαδή στο στάδιο της τελικής συνέντευξης και για λόγους στενότητας προϋπολογισμού δεν μπορούσαμε να τους χρηματοδοτήσουμε. Έρχομαι τώρα στις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας, που και αυτές είναι τμήμα της στρατηγικής του 2020 και θα ήθελα να δω πώς τοποθετείται η έρευνα στα όρια της γνώσης σε σχέση με αυτές τις ε, προκλήσεις. Αυτού του είδους η έρευνα είναι ακριβώς η έρευνα σε αυτό το οποίο δεν είναι γνωστό. Η ιστορία της επιστήμης μας έχει πει ότι πολλές φορές υπάρχουν αναπάντεχα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορεί να σχεδιάσει κανείς εκ των προτέρων και τα οποία όμως έρχονται σε αυτή την αναζήτηση στα όρια του γνωστού και του αγνώστου. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών ικανοτήτων και φυσικά παράλληλα να δίνουμε προτεραιότητα στην αριστεία στην έρευνα που βρίσκεται στα όρια της γνώσης. Εγώ πιστεύω ότι επί τη βάση του προβλεπόμενου αντίκτυπου για αυτή την έρευνα μπορεί κανείς να θέσει σαφείς στόχους, αλλά προηγουμένως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι επιστήμονες με τους οποίους εργαζόμαστε γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι ανησυχίες των κοινωνιών μας, είναι ανοιχτοί στην φωνή της κοινωνίας και, είναι ενσωματώνται αυτές οι ανησυχίες στην έρευνά τους. Για το μέλλον τώρα <clears throat> θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, επενδύουμε στους αρίστους, στους ανθρώπους που έχουν τις καλύτερες ιδέες, που εμείς τους έχουμε χρηματοδοτήσει πως αυτούς που ξεκινούν μια ερευνητική δραστηριότητα, αυτούς που εδραιώνουν και αυτούς που εκπαιδεύουν άλλους ερευνητές. Εμείς έχουμε δώσει, ε, θεσπίσει το όριο από την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μέχρι 20 χρόνια μετά από την απόκτηση του διδακτορικού είναι αυτό το οποίο λέμε ο εδρεωμένος ερευνητής. Αυτή είναι η περιοχή αυτή και τώρα θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται από 2 χρόνια ως 12 χρόνια μετά το διδακτορικό ως αυτούς οι οποίοι είναι προχωρημένοι ερευνητέ και περνούν στο στάδιο της εδραίωσης. Συζητούμε τώρα θα κάνουμε στη συνέχεια και συζητούμε Προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς θα έχουμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα έφορο κλίμα. Έχουμε διάφορους φορείς στην Ευρώπη που δημιουργούν το είδος φυτορίου όπου <clears throat> μπορεί να ανθίσει η επιστημονική δημιουργικότητα. Και θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας για τα επιστημονικά θέματα. <clears throat> Αυτά ήθελα να πω. Ας περάσω τώρα στα διοικητικά θέματα. Και εδώ πρέπει να είμαι πραγματικά ειλικρινής ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει με τόσο απλό και ομαλό τρόπο όσο θα ελπίζαμε ορισμένοι από εμάς. Έχουμε περάσει το βρεφικό στάδιο, έχουμε βγάλει δόντια και περνάμε σιγά σιγά στο πρόβλημα, στα, στην ε, πιο όρημη ηλικία. Τα προβλήματα οδοντοφυΐας όμως παραμένουν, υπήρξαν τέτοια και η μετάβαση από ένα συγκεκριμένο εφαρμοστικό φορέα μέσα στην Κομισιόν μέχρι την λειτουργία του Συμβουλίου μας ήταν κάπως οδυνηρή αυτή η μετάβαση και ένας από τους λόγους για κάτι τέτοιο είναι ότι πιστεύω ότι ένας εκτελεστικός φορέας Ε, αντιμετωπίζει τα πράγματα πολλές φορές με μονολυθικό τρόπο. Αλλά στην περίπτωση της έρευνας και ιδίως της έρευνας στα όρια του γνωστού δεν είναι αυτή μια καλή προσέγγιση. Επίσης, ο εκτολιστικός φορέας για την έρευνα έγινε κάποια στιγμή αυτόνομος, τον Ιούλιο του 2009, κάπως καθυστέρησε δηλαδή αυτή η αυτονόμησή του και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τη συγχώνευση δύο πολιτισμικών αντιμετωπίσεων, του επιστημονικού πολιτισμού που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη γραφειοκρατική κουλτούρα που βασίζεται στον έλεγχο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει βέβαια υπολογότητα και έλεγχος, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι υπήρξε μια μορφή σύγκρουσης των πολιτισμών μεταξύ των επιστημόνων και των γραφειοκρατών. Η ανάγκη λοιπόν εδραίωσης και παγιοποίησης είναι μια ανάγκη η οποία έχει γίνει αντιληπτή και ο Ιβ θα μιλήσει για την Επιτροπή Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και τα απορίσματά της. Ένας από τους λόγους όμως για όλα αυτά τα προβλήματα είναι ότι η δομή διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας έχει ορισμένες συγγενείς ανομαλίες και δυσμορφίες. Από τη μία πλευρά είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο θεσπίζει την επιστημονική στρατηγική και από αυτή την άποψη υπάρχει απόλυτη αυτονομία, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος προσπάθησε να επηρεάσει τα πορίσματα του Επιστημονικού Συμβουλίου. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει η εντύπωση ότι μπορεί κανείς να διαχωρίσει απόλυτα την επιστημονική στρατηγική από την διοικητική πλευρά. Και στην πράξη αυτό δεν λειτουργεί έτσι. Οι διοικητικές πτυχές και η επιστημονική πτυχή είναι αλληλένδετες και πρέπει να είναι αλληλένδετες πιο πολύ από ό,τι είχε προβλεφθεί στην αρχή όταν δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Επίσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι έχει επιφορτιστεί με την χάραξη της επιστημονικής στρατηγικής, δεν έχει νομικό καθεστώς, κάτι το οποίο δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα και οι σχέσεις με, την εκτελεστική, με τον εκτελεστικό φορέα και θέλω να ευχαριστήσω τον Ζακ Μικέ Υπήρξε αρμονική, αλλά <clears throat> υπήρξε αρμονική λόγω των ατόμων και όχι λόγω των δομών. Οι δομές παραμένουν έθραυστες, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα που, αυτών που καλύπτουν τις κέρδιες θέσεις. Ανακαλύψαμε επίσης ότι υπάρχει μία ε, πολύπλοκη ε, διε, διεπιφάνεια μαζί με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και δεν έχει ακόμα απλοποιηθεί και επιλυθεί το θέμα αυτό. Εμεί προσπαθούμε επομένω να ενσωματώσουμε και την επιστημονική και τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση βάσει των προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής αυτής εμείς στελεχώνουμε τώρα το φορέα μας με ένα διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο διευθυντής του εκτελεστικού φορέα, ο οποίος όμως θα είναι επιστήμον με πολύ καλή και στεναρή <clears throat> διοικητική εμπειρία. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση. Επίσης, προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε ακόμα. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε ποιο ακριβώ θα πρέπει να είναι ο ρόλο του Επιστημονικού Συμβουλίου, της, ε, ε, του εκτελεστικού φορέα. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να απλοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των εμπλοκομενων φορέων. Έχουμε εφαρμόσει άμεσα τις ε, συστάσεις της Επιτροπής Ενδιάμεσης Αναθεώσει σε σχέση με την στελέχωση με μέλη των πάνελ, που ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία είχαν δημιουργήσει προβλήματα, όπως ανέφερε και η Επιτροπή αυτή ενδιάμεσης αναθεώρηση και πιστεύω ότι προχωρούμε θετικά. Τα επόμενα τώρα βήματα που θα πρέπει να γίνουν ακολουθώντας τις συστάσεις της Επιτροπής ενδιάμεσης αναθεώρησης, όπως άφησα να εννοηθεί ήδη, είναι το πώς θα μπορέσουμε να επανακαθορίσουμε τη σχέση μεταξύ του της Γενικής Διεύθυνσης Κομισιόν, του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Φορέα. Αυτό σημαίνει να δημιουργήσουμε μόνιμες επιτροπές, να δώσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Έρευνας διευρυμένες αρμοδιότητες, να υπάρξει λοιπόν μια δυνατότητα να έχουμε επίσης πρόσβαση σε δεδομένα. Όλα αυτά είναι σημαντικά σημαντικέ ψηφίδε στο συνολικό μοσαϊκό για να μπορέσουμε εμεί να έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε σε πέρα στην εντολή μα. Και ο στόχος μας εν καιρό είναι να περάσουμε από μια κουλτούρα ελέγχου σε μια κουλτούρα αμοιβαίωτος. σε, σεβόμαστε το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε υπόλογοι, αλλά ελπίζουμε ότι στην μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανονισμών θα υπάρχει και χώρος για να μπορεί να λειτουργήσει η έρευνα στα όρια του γνωστού, να υπάρξει λοιπόν συγκεκριμένος κανονισμός εκεί, γιατί προς το παρόν εμείς λειτουργούμε επί τη βάση των συστημάτων χορήγησης που βασίζονται σε μια συμβατική βάση και δεν είναι κάτι που προσαρμόζεται με εύκολο τρόπο στις πραγματικότητες της έρευνας, ιδίως της έρευνας στα όρια του αγνώστου. Στην συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 2 Μαρτίου, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος υιοθέτησε όλες σχεδόν τις ε, συστάσεις της Ενδιάμεσης Επιτροπής, αλλά υπήρξε και ένα κενό. Υπήρξε και ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο απάντησε η Κομισιόν και αυτό ήταν κάτι το οποίο το αντιμετώπισε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος. Ζήτησε να υπάρξει μια περαιτέρω αναθεώρηση τον Ιούλιο του 2011, εφόσον θέλει ο Θεός, για να δούμε κατά πόσο τα μέτρα αυτά τα οποία έχω διαγράψει ειδοποιών σας πράγματι αποδίδουν καρπούς και αν είναι επαρκώς ικανά και ανθεκτικά να μας οδηγήσουν σε αυτήν πράγματι την ενσωμάτωση και τη συγχώνευση της διοικητικής και της επιστημονικής πλευράς όπως ανέφερα και στο παρελθόν. Όλα αυτά ανοίγουν την πόρτα για να υπάρξει μια νέα ενδιάμεσα αναθεώρηση πριν από τον Ιούλιο του 2011 η οποία θα μας επιτρέψει να δούμε κατά πόσο οι συστάσεις και οι εφαρμογές τους έχουν πράγματι προσαρμοστεί επαρκώς στην ανάγκη να πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας την απαραίτητη για αυτό δομή. Ατενίζω τώρα επέκεινα του προγράμματος έρευνας 7 είναι ελπίς ότι το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας θα είναι ένας μόνιμος οργανισμός. Προς το παρόν εμείς βρισκόμαστε μέσα στο χρονικό ορίζοντα του 7ου προγράμματος πλαίσιου μέχρι το 2013. Θα θέλαμε να δώσουμε μια μόνιμη μορφή σε αυτό το φορέα, ένα ιδιότυπο σου generis ε, όργανο με ειδικό προϋπολογισμό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα καθήκοντά του και νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα επανακαθορισμό αρμοδιοτήτων και λειτουργίας εφόσον απαιτείται κάτι τέτοιο και θα ήθελα να κλείσω εδώ και να σας ευχαριστήσω όλους για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο αναλυτική σας παρουσίαση. Θα έλεγα να ακούσουμε πρώτα και τους τρεις ε, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Παρακαλώ, κύριος Μένι έχει το λόγο. Πρόεδρε, μέλι, αγαπητό μέλη, θα ήθελα να σας πω ποια ήταν η δική μου εμπειρία ως εισηγητή σε αυτήν την Επιτροπή. Θα πρέπει να σας πω ότι όταν συστάθηκε το ERC ήμουν κάπως σκεπτικός για αυτό τον οργανισμό γιατί θεώρησα ότι μία ενδυνάμη αδυναμία θα έγκυτο στην αξιολόγηση, στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Και ήμουνα σκεπτικός, διότι είχε σημασία τι συνέβη σε άλλα προγράμματα της Κομισιόν όπου η διαδικασία αξιολόγησης μερικές φορές δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Επίσης, κλήθηκα να είμαι εισηγητής σε αυτήν την Επιτροπή, διότι όταν ήμουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο συμμετείχα στην όλη διαδικασία, διαθεσμική διαδικασία. Σήμερα είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος και εκφράζω τις ε, προσωπικές μου απόψεις και τις ε, απόψεις της Επιτροπής και δεν θα αποκρύψω τίποτα γιατί θα φοβόμουν ότι θα μπορούσα να ζημιώσω ε, έναν φορέα ή θεσμό. Μετά από μήνες ερευνών και ανάλυσης με βάση ακροάσεις, έρευνες και την τεκμηρίωση που διαθέτουμε, στα πλαίσια της Επιτροπής φτάσαμε σε ορισμένα σαφή συμπεράσματα. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία και είναι το διαμάντι στην κορώνα της έρευνας που, όπου ο μεγάλος χορηγός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν πρόκειται να επέλθουν βελτιώσεις θα μπορέσουν να σταθούν ως ένας φάρος για άλλα προγράμματα τα οποία θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Άρα αυτή η επιτυχία είναι σαφής, είναι ευκρινής. Ακριβώς επειδή πολύ αφοσίωσαν, αφιέρωσαν το χρόνο τους για το εγχείρημα αυτό. Καταρχήν η επιστημονική κοινότητα καθε αυτή. Είχαμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο Ήταν ένα πολύ ε, καλό πρόγραμμα μεταξύ των εθνικών και των διεθνών προγραμμάτων που επέτρεψε στους επιστήμονες να συνεργαστούν κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω τεχνητό. Δηλαδή, τις πρωτοβουλίε τις αναλάμβαναν με μονομένα άτομα και οι ομάδες τους. Επρόκειτο για μία ε, δίκαιη, σωστή διαδικασία αξιολόγησης. Και επειδή είχαμε να κάνουμε με μία ε, συγκεκριμένη διάρθρωση στην οποία είχαμε, η οποία μας είχε απασχολήσει, απέδωσε, υπήρξε ένα θαύμα, έτσι ώστε να καταπραϊνθούν οι δυσκολίες τις οποίες θα αναφερθώ. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι παρά από αυτή την επιτυχία υπήρξε ε, μεγάλη απογοήτευση για όχι εύλογους λόγους. Δηλαδή, αν ζητήσετε από έναν αναθεωρητή να αποδείξει την ταυτότητά του και την ίδια του την ύπαρξη και να συμπληρώσει πολλές ε, διατυπώσεις και φόρμες χωρίς να πληρωθεί, γιατί θα πρέπει να το κάνει. Γιατί εργάζεται αμισθή και του επιβάλλεται ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες είναι καθαρά γραφειοκρατικές ε, ως προς τον τύπο και την ουσία. Αυτό φαίνεται κάτι το καθαρά κοσμικό, όμως δεν είναι. Γιατί ένα σύστημα αξιολόγησης της έρευνας αφορά την ποιότητα των αξιολογητών. Άρα οι αξιολογητές θα πρέπει να είναι καλύτεροι από τους προτείνοντες. Διαφορετικά είναι παράλογη η διαδικασία. Για να έχουμε τους καλύτερους αναθεωρητές θα πρέπει να τους πείσουμε ότι εργάζονται ως καλοί πολίτες της επιστημονικής κοινότητας ακόμα και εάν εργάζονται αμυστοί. Και μπορώ να σας πω Διαβάζοντας τα σχόλια ιδιαίτερα των μη Ευρωπαίων επιστημόνων για τον τρόπο που λειτουργήσε η Κομισιόν ε, ως προς αναθεωρήσεις ήταν ε, κάτι το τρομακτικό. Επίσης υπήρξε ανεπαρκής διάρθρωση. Είχατε την, ε, τον Γενικό Γραμματέα της ΙΑΣΕ και μετά είχατε τον ε, γραμματέα της διάρθρωσης εφαρμογής. Δεν ήταν καλοί ή κακοί ή δεν ήθελαν να συνεργαστούν. Και εάν ήταν λειτουργικό το σύστημα είναι επειδή συνεργάστηκαν. Αλλά για διαρθρωτικούς λόγους δεν λειτουργήσε καλώς το σύστημα. Γι' αυτό ζητήσαμε να συγχωνεύσουμε αυτές τις δύο λειτουργίες. Δεν αρκεί αυτό έτσι ώστε αυτή η αναθεώρηση, η μεταρρύθμιση να είναι επιτυχής. Αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν αυξητικό, μπορώ να πω, τρόπο λειτουργίας και όχι έναν ριζοσπατιστικό, ε, ξεκινώντας από το μηδέν. Γιατί ξέρετε, χρειάζονται δύο-τρία χρόνια συζητήσεων πριν ληφθεί μία απόφαση. Άρα επιλέξαμε έναν λογικό δρόμο αλλά η επιτυχία αυτής της μεταρρύθμισης δεν αφορά τις νέες ε, διαρθρώσεις, αλλά το πνεύμα που θα μας ε, διέπει. Τέλος, είμαστε πεπισμένοι ότι επρόκειτο για μία επιτυχία, αλλά ήταν ε, ευάλωτο το οικοδόμημα. Και αυτό σχετίζεται ε, με το γεγονός ότι ε, ο, ως, έγκυται στη διαφορά μεταξύ μέσων και αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μεταξύ έρευνας και καινοτόμου έρευνας και μπορούμε να πούμε ότι ως προς αυτό τα διοικητικά μέσα ήταν γραφειοκρατικά και μη ευκίνητα. Θα πρέπει να άρουμε τέτοιες αντιφάσεις στο μέλλον. Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι προσωπικό. Σας είπα ότι θα είμαι ειλικρινής. Το ERC, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, δεν αποτελεί εξαίρεση στο, στον κανόνα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι η καλύτερη περίπτωση μιας κατάστασης που δεν είναι ικανοποιητική, διότι υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία στην όλη διαδικασία. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς διότι βασίζονται στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Φαίνεται ότι όλοι είμαστε εγκληματίες, πρέπει να μας ελέγχουν, να μας εποπτεύουν και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε για ε, έναν πολιτισμό της αξιολόγησης όπως ισχύει στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Εμένα με ελέγχουν 10-20 φορές κάθε χρόνο. Αλλά δεν με αποτιμούν ως ε, επιστημονικό οργανισμό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να ε, επιλέξουμε έναν ιεραρχικό τρόπο μετασχηματισμού να δούμε ποιες ήταν, ποια ήταν η αξία του ΕΣΕ. Ε, υπήρχε αυτονομία και δεν υπήρχε συνάφεια με τις χρηματοδοτικές προτάσεις. Άρα θα συγχωνεύσουμε την Γενική Γραμματεία και την ε, Γενική Διεύθυνση των ε, οργανισμών αυτών, των εκτελεστικών οργανισμών. Θα πρέπει επίσης να ορίσουμε ένα αναγνωρίσιμο ε, επιστημονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να βρούμε έναν πολύ καλό διοικητή. Διότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη με το κατεστημένο της Κομισιόν. Επίσης, οι κανονισμοί θα πρέπει να είναι πιο φιλικοί προς το χρήστη, ιδιαίτερα ως προς τα μέλη του πάνελ που δουλεύουν ε, αμυστή, διότι αυτό είναι το ζωτικό σημείο για να διασφαλίσουμε την ποιότητα αυτού του νέου ε, φορέ. Επίσης θα πρέπει να αναθερούσουμε τη διαδικασία επιλογής των μελών του πάνελ και των αξιολογητών μέσα από μία δημόσια τράπεζα δεδομένων. Θα πρέπει να δούμε την ε, διαδικασία συμβάσεων και αυτό με βάση καταποκοπήν ποσά. Διότι το σύστημα χρηματοδότησης μέσω συμβάσεων είναι ένα παράλογο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να μετατραπεί σε ε, συγκεκριμένα ε, καταποκοπή ποσά και διαδικασίες. Να μην μιλάμε για έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεχής ελέγχους, διότι ε, η ζωή μας είναι, η επιβίωσή μας είναι αδύνατη σε επίπεδο κομισιών. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν υποβάλλουν προτάσεις εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και είναι ένα παράδοξο να είμαστε τόσο παθητικοί σε ακαδημαϊκό επίπεδο τη στιγμή που ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ένας γενναιόδωρος ε, πάροχος και χρηματοδότης. Άρα για το μέλλον ας ελπίσουμε καταρχήν να εφαρμοστεί αυτή η έκθεση. Είμαι πεπισμένος για κάτι τέτοιο και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής προς τον κύριο Ποτότσνικ, τον πρώην Επίτροπο Έρευνας. Επίσης χαίρομαι διότι θα γίνει μια αξιολόγηση σε δύο χρόνια γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το φορέα να μετατραπεί σε μια ρουτίνα. Θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός να δίνει συγκεκριμένες οθήσεις και να ε, δέχεται οθήσεις. ας ε, προβάλλουμε αυτή την αυξητική στρατηγική, incremental strategy. Αν όμως δεν είναι λειτουργική, ας ε, προχωρήσουμε πέραν αυτής, διότι χρειαζόμαστε ε, ο οργανισμούς που να παρομοιάζουν με τους ε, αμερικανικούς οργανισμούς. Ο Έλια Ζερουνί είναι ένας επιστήμονας αλγερινής καταγωγής, ε, ε γαλλικής, ε, ε, γαλλικού πολιτιστικού υποβάθρου, ο οποίος διέπρεψε στην Αμερική. Ήταν ε, επικεφαλής ενός φορέα που ήταν ε, κατά 20 φορές πλουσιότερος από τον ΕΣΕ και δεν πίστευε στα μάτια του όταν διάβαζε για αυτόν τον οργανισμό. Ήταν όμως πεπισμένος ότι η, η Ευρώπη θα πρέπει να έχει έναν αντίστοιχο φορέα, επιστημονικό οργανισμό. Και ο διάβολος βέβαια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, όπως λένε οι Βρετανοί μας φίλοι. Θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους, μπορούμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση. Αν δεν έχουμε την, την κατάλληλη οργάνωση, θα αποτύχουμε. Άρα τώρα ε, ένας εκτελεκτιστικός φορέας ε, διοικεί το ΕΣΕ Γι' αυτό θα πρέπει να είναι αρκετά ε, αυτόνομη. Εάν αυτός ο εκτελεστικός φορέας υπηρετεί μια μεγαλύτερη γραφειοκρατία, τότε ξεχάστε το. Δεν θα επιτύχει σε αυτό που όλοι επιθυμούμε για το ΕΣΕ. Δηλαδή να τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης. επειδή βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό φορέα και έχουμε εκλεγεί για μια περιορισμένη θητεία, θα ήθελα να εκφράσω μία επιθυμία, δηλαδή να προωθήσουμε την έρευνα όχι αύριο αλλά στο εγγύς μέλλον. Παρόμοιοι οργανισμοί χρειάζονται χρόνο και περισσότερες από μία θητεία έτσι ώστε να αποκτήσουν ε, σώμα και σκοπό. Θα πρέπει να είναι ένας φάρος ο οποίος να μας καθοδηγήσει στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξετε αυτό το φορέο για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Διότι όταν μιλάμε για έρευνα Μιλάμε για ένα μακροχρόνιο πλαίσιο, ε, επενδυτικό πλαίσιο καταρχήν και είμαι πεπισμένος ότι τώρα που δημιουργήθηκε αυτός ο, ο φορέας μπορεί να λειτουργήσει σωστά για το μέλλον. Ευχαριστώ για την Πολύ σαφή αυτή η παρουσίασή σας, αλλά πολύ χρήσιμη στην συζήτησή μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα εμπλουτίσετε έτσι την συζήτησή μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μέτη, να μας κάνει τη δική του παρουσίαση. Και μετά οι συνάδελφοι θα μπορούν να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Μέτη, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να βρω εδώ την παρουσίασή μου στον υπολογιστή. Maybe we need some help from your assistant. Ίσως κάποιος να μπορεί να με βοηθήσει εδώ. Yeah, yeah I'm trying to. Sometimes there are problems that only for and problems are there to be solved. Super. Okay. Merci. Well, good afternoon to everybody. It's a pleasure to be... Καλησπέρα σας. Ε, είναι πολύ μεγάλη ευχαριστησή μου να είμαι εδώ για διάφορους λόγους. Καταρχήν γιατί το Κοινοβούλιο ε, συνέβαλε στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα, ε, του ΕΣΕ, ήταν ένα στοιχείο στην απόφαση. Ψήφισε επίση η δημιουργία τη Εκτελεστική Επιτροπή. Θυμάμαι την ψηφοφορία αυτή από μερικά χρόνια και είμαστε και υπόλογοι στο Κοινοβούλιο που είναι η Δημοσιονομική Αρχή και επίσης είμαστε υπόλογοι και για τον διοικητικό, το, το διοικητικό τμήμα. Άμεσα υπόλογοι λοιπόν. Έχω να σας περάσω κάποια μηνύματα. Καταρχήν θα ήθελα όπως και συνάδελφοι έτσι και εγώ να σας πω ότι είναι επιτυχής η ιστορία του ΕΣΕ, μια πολύ καλή αρχή συνεχίζεται. Σαν αρχή πάντως είναι καταπληκτικό. Δεύτερον, να σας πω ότι ως δομή χρησιμοποιούμε μια χρηματοδότηση σημαντική 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό μέσω της ε, υπηρεσίας μας το κάνουμε πιο φτηνά και γρήγορα. Και το τρίτο σημείο είναι ότι η δομή του ΕΣΕ είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να δούμε καταρχήν ε, πώς λειτουργεί η ΕΣΕ και να δώσω κάποια παραδείγματα. Είναι κάπως νωρίς ίσως γι' αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε κάποια πολύ επιτυχή αποτελέσματα. Θα πω δύο λόγια για το πώς η Επιτροπή και η, η υπηρεσία μας ακολουθεί τις συστάσεις ε, του πάνελ αναθεώρησης και να σας υπενθυμίσω τους κυρίους στόχους για την Ευρώπη για το 2010. Το πρώτο είναι να σας πω ότι πρόκειται για μια νομική οντότητα Γι' αυτό αρχίζω με αυτό τον ε, πίνακα εδώ. Βασιζόμαστε στα άτομα που μας εκπροσωπούν. Όλοι αυτοί είναι κατά βάση κρατικοί υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στο ΕΣΕ. Εδώ βλέπετε μια κατανομή του προσωπικού μας ανάλογα με την ε, υπηκότητά τους. Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας έχουμε πλήρη πολυεθνικότητα στο ε, προσωπικό μας, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να καλύψουμε τις διάφορες ε, πολιτιστικές ε, τάσεις Ευρώπης. Επίσης, είμαστε πολύ περήφανοι να σας δούμε ότι τα δύο τρίτα του προσωπικού είναι γυναίκες, μόνο το ένα τρίτο είναι άντρες, εν αντιθέσει προς άλλες υπηρεσίες και όσον αφορά τους επισυμβάσει υπαλλήλου σε πολύ ψηλό επίπεδο πάντα. Βλέπετε στον πίνακα αυτό ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό των λεγόμενων Research Program Officers, δηλαδή υπαλλήλου τους ε, ε, για τα ερευνητικά προγράμματα, 35 ε, άτομα με διδακτορικό Εδώ βλέπετε την εξέλιξη του προσωπικού. Αρχίσαμε πραγματικά από το μηδέν. Και βλέπετε ότι γλίγορα μπορέσαμε Έχουμε 287 άτομα που εργάζονται σε μας, μικρό το μέγεθος, αλλά το μέγιστο θα είναι 389 το 2013. Σε αυτή την γραφική παράσταση βλέπετε ότι και κάτι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι είναι υπάλληλοι επισυμβάση που εργάζονται για διοικητικά θέματα και μας υποστηρίζουν ενώ οι προσωρινοί πάλι ασχολούνται με τα επιστημονικά θέματα. Όσον αφορά το, το διοικητικό προϋπολογισμό, αυτό ενδιαφέρει πολύ το Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρος. Εμείς διαφοροποιούμε από τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε κάτω του 3,5% του, διοικητικού μας του λειτουργικού μας κόστος για τη διοίκηση. Και η Ξεκονομήσεις που κάναμε από τη διοίκηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για έρευνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτόν τον πίνακα είναι ότι μισθή, επιδόματα κατοιχείας ε, ε, και πληροφορική είναι το 85% των δαπανών μας. Ε, φυσικό είναι αυτό. Τώρα, εξτάζω στην διαδικασία αξιολόγησης. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ε, επιλέγει τους ε, επιστήμονες που θα εργαστούν σε εμά. Και δεν είναι μόνο υψηλού επίπεδου, υψηλού όγκου επίσης. Έχουμε περίπου 3.000 προτάσεις για κάθε ε, διαγωνισμό. Έχουμε αξιολογήσει 9.000 περίπου σε τρία χρόνια. 19.000 σε τρία χρόνια. Και περαιτέρω ε, καταφέραμε να ολούσουμε χίλια άτομα στα πάνελ, που είναι πάρα πολύ αξιολογή πηγή αυτό, γιατί εξαρτάται η αξιοπιστία μας από το πόσο καλό είναι το σύστημα αξιολόγησης και επίσης έχουμε και άλλους χίλιους συμπραγματικούς λεγόμενους αξιολογητές εξ αποστάσεως ε, για κάθε διαγωνισμό. Όπως σας είπα, τα μέλη αυτών των πάνελ ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και μπορούμε να προσελκύσουμε άτομα από όλο τον κόσμο, 10% παραδείγματος χάρη, είναι από χώρες εκτός Ευρώπης. Και υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, γιατί υπάρχει κάποια ειδωτερότητα έτσι, και δείχνουμε ότι το ΕΣΕ είναι πολύ καλά συνδεδεμένα με τα καλύτερα ευνητικά συστήματα και προγράμματα του κόσμου. Και παρεμπιπτόντω, πολλά από τα μέλη πάνελ έχουν πάρει βραβείο Νόμπελ που βλέπετε πόσο ενδιαφέρονται για την εργασία μας. Ακόμα εξίσου ενδιαφέρον είναι, εξετάζοντα την αξιολόγηση των απολυσμάτων, ότι 10 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμο, προσαρτίζονται. Δηλαδή, εάν εμεί βρούμε κάποια άτομα ιδιαίτερα αξιόλογα, οι χώρες αυτές χρηματοδοτούν, αν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, τους εν Και επίσης έχουμε και κάποια κράτη-μέλη που έχουν ε, παρόμοια συστήματα σήμερα. Παραδείγματο χάρη θέλω να αναφέρω εδώ την Πολωνία. Για να έχετε μια ιδέα τι τύπου αναλύσει μπορούν να γίνουν από τα αποτελέσματά μα. είναι παραδείγματο χάρη επιδοτήσει για αρχάριου ε, ερευνητέ. και επίση ε, για την πρόθεση της κινητικότητας. Στο αριστερό τμήμα του πίνακα έχετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το Ηνωμένο Βασίλειο Φερρυπίν. όπου αυτό που είναι σαν τη γαλλική σημαία, μπλε, άσπρο, κόκκινο, είναι υπήκοοι εκτός του Ευρωπαϊκού, του Ηνωμένου Βασιλείου, συγγνώμη, που έχουν προσελκυστεί να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το, το καθετή τμήμα είναι η υπήκοή του Ηνωμένου Βασιλείου. Και προς τα μέση βλέπετε την Ελβετία που επίσης μπορεί να προσελκύσει πάρα πολλούς εκτός της χώρας αυτής. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το τμήμα του μπλε. Εν αντιθέσει με αυτό βλέπετε το Βέλγιο που είναι κατά βάση όλοι Βέλγοι. Αλλά από μια τέτοια ανάλυση θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ε, ερευνητική πολιτική, γιατί είναι θαυμάσια άτομα όλοι αυτοί. Και αν δείτε πόσο ελκυστικά είναι, βλέπετε στην εικόνα αυτή τον αριθμό των υποψηφίων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πέντε παραδείγματος χάρη άτομα έρχονται εκτός Ευρώπης από την Ιαπωνία αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ε, μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε εκείνους που προέρχονται από την Ευρώπη και επανέρχονται, ιδίως από τη ΣΥΠΑ. Θα θέλαμε να προσελκύσουμε και πραγματικούς Αμερικανούς, αλλά και άτομα από αναπτυσσόμενες χώρες, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και άλλες. Ορισμένα σημαντικά στοιχεία, προπολογισμό για το 2010 είναι 1,2 δισεκατομμύρια, μεγαλύτερο κονδύλιο στην Γενική Διεύθυνση Έρευνα που αυξάνεται ε, κατά 250 εκατομμύρια ανά έτος. Ήδη 900 χορηγήσεις έχουν υπογραφεί, ο ρυθμός θα αυξηθεί. Και τώρα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τους δείκτες απόδοσης. για να τα συγκρίνουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε τον Εθνικό ε, το Εθνικό Δήμα Έρευνα στι Πολιτείε, όπου 70% των ετούντων γνωρίζουν για το αποτέλεσμα των αιτήσεών του μέσα σε 6 μήνε. Το να υπάρχουν ε, απαντήσει γρήγορα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε λοιπόν τον Αμερικανικό φορέα και βλέπετε τι έχει γίνει στη δική μα περίπτωση. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο του NSF στην Αμερική, αλλά πλησιάζουμε. Δηλαδή, Είμαστε στο ίδιο γήπεδο ακόμα και έχουμε επομένως ενδείξεις ότι τα πράγματα λειτουργούν καλά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ο χρόνος μέχρι την καταβολή της πληρωμής που δημιουργεί, σε πολλές, δημιουργεί πολλές προστριβές πολλές φορές στον ερευνητικό χώρο. Εμείς πληρώνουμε το 100% εγκαίρος, όχι μονάχα οι προπληρωμές αλλά και οι ενδιάμεσες πληρωμές. Βλέπετε ποιος είναι ο, ο μέσος χρόνος, 15 και 20 μέρες και αυτό οδηγεί σε μια ικανοποίηση για την ε, διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Έρευνας. Ο κύριος Μίνη ανέφερε τη δυσκολία που είχαμε <clears throat> με τους ε, αξιολογητές. Δεν ήταν σπάνιο να έρχονται αξιολογητές από τις ΗΠΑ και να χρειάζονται να περάσουν μήνες για να καταβληθούν οι αμοιβέ τους. Από τότε που εμείς είμαστε αυτόνομοι, έχουμε καταφέρει να γίνεται αυτή η αποπληρωμή μέσα σε 17 μέρες κατά μέσον όρο. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική βελτίωση. Τώρα, κάποια παραδείγματα για να σας δείξουμε τι κάνουμε. παίρνω δύο σχέδια στον τομέα της ενέργειας που είναι πολύ σημαντική πρόκληση για όλους μας. Καταρχήν τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, η φωτοβολταϊκή ενέργεια. Ξέρετε ότι η μεγάλη δυσκολία εκεί είναι το να αυξήσει κανείς την ε, αποδοτικότητα των ημιαγωγών. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ε, ημιαγωγοί που χρησιμοποιούν και την ε, μεταφορά φορτίου και την συλλογή φωτός ο στόχος είναι να υπάρξει μια αποδέσμευση αυτών των δύο δραστηριοτήτων και αυτό θα μας οδηγήσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την κβαντική αποδοτικότητα στα 11 με 15%. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Ένα δεύτερο αφορά τη χρήση υδρογόνου ως ε, καυσίμου για οχήματα. Είναι δύσκολο να παραγάγει κανείς και να αποθηκεύσει το υδρογόνο όπως γνωρίζετε και στις διαδικασίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούμε ορισμένε χημικές ουσίες. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο εκτελείται στο Ισραήλ χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιεί αυτούς τους χημικούς παράγοντες μαζί με φως και επομένως έχει μεγάλη αποδοτικότητα ενέργειας. Τώρα το θέμα των αναθεωρήσεων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα και έρχομαι στο θέμα αυτό πιο λεπτομεριακά γιατί ήδη έχει αναφερθεί πολύ κλήρο στο θέμα των συστάσεων της ενδιάμεσης αυτής μεταρρύθμισης, αλλά και η Κομισιόν και φυσικά και ο εκτελεστικός φορέας υπογραμμίζουν τη σημασία της ποιότητας αυτού του έργου, αυτής της ε, ενδιάμεσης ε, <clears throat> αναθεώρησης και του Προέδρου και όλης της ομάδας αυτής και από την ε, έκθεση αυτή για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Εμείς εκδώσαμε μια ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 2009, όπου υπάρχει ο δικός χάρτης για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να γίνουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται δύο χρόνια για να επιτευχθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και το ανέφερε εδώ και η Έλγα. Επομένως, γενικά έχουμε ένα σημείο συνάντηση τον Ιούλιο του 2011 για όλα αυτά, όλες αυτές τις ενέργειες. Τα κύρια θέματα τώρα τα οποία γίνονται. Πρώτα απ' όλα το θέμα της διακυβέρνησης όπως αναφέρθηκε ότι έχει ένα χαρακτήρα ροκοκό η διακυβέρνηση. Να μπορέσουμε να συγχωνεύσουμε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ΕΡΣΕΑ και του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Να υπάρξει ένα άτομο λοιπόν και μόνο το οποίο θα είναι ένας διακεκριμένος ε, επιστήμονας με πολύ καλή διοικητική εμπειρία. Αυτό είναι και η οικονομία αν θέλετε. Βελτίωση δεύτερον της, των διοικητικών διαδικασιών, παραγωγικά, χάρη σε ό,τι αφορά την απόδοση εξόδων των εμπειρογνωμόνων και τρίτον η πιο επαγγελματική μορφή των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύστημα υποστήριξη στα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που αυτή τη στιγμή εργάζονται περίπου σε φιλανθρωπικό επίπεδο, αλλά είναι πάρα πολλή εργασία που πρέπει να φέρουν σε πέρα. Πρέπει να δημιουργήσουμε επίση και μία ανεξάρτητη επιτροπή ταυτοποίηση για, για τα άτομα τα οποία θα αναλάβουν την ε, ανανέωση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Αυτό είναι μια ενεξελίξη ακόμα διαδικασία και επίση θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δράσει του Συμβουλίου θα είναι πιο διάφανε σε σχέση με του εξωτερικού εμπλεκόμενου. Δηλαδή τα πρακτικά μα να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Χρονοδιάγραμμα. Ο διευθυντή πρέπει να, να διοριστεί στα μέσα του 2010 νέες διαδικασίες για τους εμπειρογνώμονες και την απόδοση εξόδων περατώνονται τώρα, οπότε έχουμε προχωρήσει αρκετά στον τομέα αυτό. Όπως είπε και ο Ιβ πολύ καλά, η κουλτούρα σε ό,τι αφορά τα ρυθμιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα, τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καλά προσαρμοσμένη στην έρευνα στα όρια της γνώσης. Χρειάζεται μια απλοποίηση της χρηματοδότησης, απλές διαδικασίες δηλαδή, για να εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει σωστή διαχείριση, ε, καλύτερη απλοποίηση και το υπόλογο, ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και του ελέγχου και πιο αποτελεσματικό εκτελεστικό φορέα. Αλλά γενικά είναι θετικά τα πράγματα για την εφαρμογή των προγραμμάτων μα. Το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα βέβαια δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα, είναι πια ένα θεσμό. Και εδώ τίθεται το θέμα τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού βάσει μια πρόταση που θα προέρχεται από την Κομισιόν τον Ιούνιο του 2010. Τελευταία διαφάνεια, το 2010. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα λάβουν χώρα. Ανάπτυξη της επιστημονικής μας στρατηγικής, του Επιστημονικού Συμβουλίου για να έχουμε μεγαλύτερη ακτινοβολία και σε άλλες χώρες του κόσμου πέραν της Ευρώπης, να έχουμε νέα εργαλεία, να έχουμε καλύτερες σχέσεις με εθνικούς φορείς χρηματοδότησης, να λειτουργήσει λοιπόν η επικουρικότητα και να δώσουμε επίσης και έμφαση στο τομέα της καινοτομίας και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία του επομένου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα η δεύτερη φάση της εφαρμογή του Συμβουλίου. Και εδώ είναι σημαντική, είναι αυτά που είπα προηγουμένω και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα θέλουμε να εμπλακεί και το Κοινοβούλιο, θα γιορτάσουμε το χίλιο στο τη χιλιοστή χορήγησή μας και κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας θα ξεκινήσει και η... θα γίνει και μια τελετή για την ε, ε, απόδοση των χορηγήσεων σε αυτούς που ξεκινούν την έρευνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, και ο Πρόεδρος. Έστω λιγάκι γιατί στις 6 έχουμε πάλι ένα, ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα να δώσω τους συναδέλφους ε, τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις αν θέλουν. Λοιπόν, καμία μακρά εισαγωγή. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Α, έχω τον κατάλογο, συγγνώμη. Ο κύριος Καλάς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για δύο λόγους, όχι μόνο γιατί μου δίνετε το λόγο, αλλά και γιατί με ευχαρίστηση βλέπω ότι ο προγραμματισμός που είχατε κάνει από τον παρελθόντα Σεπτέμβριο και είχατε υποσχεθεί ότι ζητήματα έρευνας θα έρχονται συχνότερα σε αυτή την Επιτροπή, ακολουθείτε και είναι μεγάλη μου η χαρά που έτσι γίνεται. Μεγάλη χαρά έχω επίσης επειδή συναντώ την κυρία Νοβότνη ως καθηγήτρια. Την είχα συναντήσει ως μέλος του ERC στο παρελθόν και τώρα τη βρίσκω πρόεδρο. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Εκείνο τον καιρό υπηρετούσα ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας της χώρας μου και είχα την ευκαιρία <clears throat> να παρακολουθήσω τη γέννηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ERC. Θέλω να ευχαριστήσω τους άλλους δύο κυρίους να συμφωνήσω με τον κύριο Χένι ότι θα ήταν αδικία να μην μνημονεύσουμε το έργο του κυρίου Ποτόσνικ, ο οποίος πρακτικός προσπάθησε να κάνει αυτό που αποτύχαμε να κάνουμε στην οικονομική πολιτική, δηλαδή να δώσει ενιαίο στίγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από την ΕΡΑ, την κινητικότητα των ερευνητών, το ERC, τις υποδομές στο ΕΣΦΡΙ, τους μεγάλους οργανισμούς με τη δυνατότητα που έχουν να κάνουν big science, όπως είναι το CERN, όπως είναι η ESA, όπως είναι το GRC. Ε, Ήταν επιτεύγματα του κυρίου Ποτόσνικ, τον οποίον και εγώ ευγνωμονώ, διότι έδωσε άλλη διάσταση που μέχρι τότε δεν υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο όραμα της ερευνητικής της πρωτοπορίας. Όμως, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρεί εν κενό, προχωρεί μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και τα βήματά της δεν μου φαίνεται να ανταποκρίνονται ούτε στις προοπτικές του 2025, όπως η ίδια με τη μελέτη που έκαμε a με τη μελέτη των Αμερικανών, δηλαδή Trends in 2025, δεν μου φαίνεται να μπορούμε για την ώρα να ισχυριστούμε όπως ο κύριος Μέθεϊ είπε, ότι είμαστε κοντά με το NSF. Θα ήταν νομίζω αυταπάτη να πούμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε ένα σύστημα όπως είναι το αμερικάνικο, όπου το τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή η ε, εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, λειτουργούν εδώ και 50 χρόνια με μεγάλη και πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη δική μας. Είχα την ευκαιρία σε άλλες παρεμβάσεις μου να πω ότι είναι κρίμα που η Ευρώπη ύστερα από 400, 400 χρόνια επιστημονικής ηγεμονίας φαίνεται από το 1950 και μετά να μην μπορεί να ακολουθήσει τα ίδια βήματα. Είμαστε πάντα κοντά, αλλά όχι και ποτέ πρώτοι. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως την διαφορετική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ένα κάτι τύπου οι Αμερικάνοι το κάνουν πριν από πολλά χρόνια. Άρα τώρα ο διεθνής ανταγωνισμός απειλεί όχι μόνο εμάς, απειλεί και την Αμερική. Είμαστε χαρούμενοι για το EIT, την ίδια ώρα που στην Ινδία έχουν κάνει 12 EIT είμαστε χαρούμενοι και λέμε ότι ε, έχουμε πολύ καλά επιστημονικά αποτελέσματα. Το συνολικό επιστημονικό παγκόσμιο αποτέλεσμα εξακολουθεί να γέρνει υπέρ της Αμερικής. Το ίδιο σημαίνει με τις πατέντες, το ίδιο συμβαίνει και με την big science. Η γραφειοκρατία πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας δεν συμβαδίζει, ταπεινώνει και είναι εκτός στόχου της υψηλής επιλεκτικότητας που σοφά εφαρμόζει το Επιστημονικό Συμβούλιο και το EIT. Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνετε ανθρώπους με γραφειοκρατίες που έχουν ως ένδειξη ότι θεωρούνται απαταιώνες εκ προημίου όταν επιχειρείτε να συλλέξετε τους άριστους. Αυτά δεν συμβαδίζουν. Τέλος, είχαμε σήμερα κύριε Πρόεδρε την ευκαιρία να ακούσουμε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι τόνισαν δύο πράγματα. Την ταπείνωση της Ευρώπης από την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, αποτυχία η οποία συνοδεύει και τα οράματα για το 2020 και τέλος ως φάρμακο για αυτήν την κατάσταση τους ακούσαμε να προτείνουν επικέντρωση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι πράγματι μόνο αυτή η μέθοδος μπορεί να μας σώσει, να μας λυτρώσει και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε παρά μόνο ένα δρόμο. Όχι μέτρα συνοχής εκεί που χρειάζεται ανταγωνιστικότητα. Μας το έδωσε γραμμένο και η, Σουηδική Προεδρία. Σκληρός ανταγωνισμός για να βρούμε τους άριστους. Είμαι από μια χώρα που δεν με συμφέρει να το λέω, όμως αισθάνομαι πρώτα Ευρωπαίος και συνεπώς το καθήκον της Ευρώπης είναι αυτό. Για το λόγο αυτό έχω να συγχαρώ την κυρία και τους κυρίους για το σπουδαίο έργο που ε, κάνουν και εσάς κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλάμε για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου και τον κύριο Ματέη, θέλω να τον ευχαριστήσω όλους για το έργο που έχουν φέρει σε πέρας μέχρι τώρα για την εφαρμογή του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος, το οποίο υποστηρίζει την έρευνα στα όρια μέσα στα τωρινά πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα τώρα μία πιο διοικητικού χαρακτήρα και μία σε σχέση με την μορφή που θα έχει το μέλλον. Η διοικητική ερώτηση είναι αν έχετε διερευνήσει όλες τις δυνατότητες για την απλοποίηση των κανόνων. Το θέτω αυτό το ερώτημα γιατί παρακολουθώ από πολύ κοντά και το Ευρωπαϊκό Ένδρυμα Τεχνολογίας από τα γενοφάσκε του και πιστεύω ότι κατάφεραν, ίσως γιατί χρησιμοποίησαν και τις προηγούμενες εμπειρίες σας, έχουν καταφέρει μέσα στο δημοσιονομικό κανονισμό που έχουμε ακόμα να προχωρήσουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά την απλοποίηση αλλά, των κανόνων, αλλά και σε ό,τι αφορά την αυτονομία τους. Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο Τεχνολογία Τεχνολογίας έχει μεγαλύτερη αυτονομία από ό,τι η Επιστημονική Επιτροπή σας. Προβλέπετε λοιπόν <clears throat> να υπάρξει κάποια διαρρεύνση περαιτέρω δυνατοτήτων ή περιμένετε να υπάρξουν ριζικέ αλλαγέ προηγουμένω στο δημοσιονομικό κανονισμό για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε περαιτέρω απλοποίηση. Το δεύτερο ερώτημα αφορά περισσότερο την ουσία, δηλαδή τη μορφή που θα έχει η έρευνα στο μέλλον και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένω. Γυρωμένη. Είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα ω μοχλού αλλαγή, καταλήτη αλλαγή, αν θέλετε, στο ευρωπαϊκό στερέωμα έρευνα. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο είναι κατεπήγον να υπάρχει μια κοινή επιλογή προτάσεων. Είπατε ότι το κάνετε αυτό ήδη σε επίπεδο άτυπο, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη επιλέγουν, επιλέγουν επί εθελοντικής βάσης προτάσεις και χρηματοδοτούν προτάσεις που εσείς δεν είχατε αρκετά λεφτά να χρηματοδοτήσετε. Βλέπετε κάποια δυνατότητα να υπάρξει λοιπόν αυτή η κοινή δράση με τα κράτη-μέλη, συζητάτε στο Επιστημονικό Συμβούλιο τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να θεσμοποιηθεί περισσότερο αυτή η άτυπη συνεργασία και με ποιο τρόπο θα συμβάλλεται στο να υπάρχουν κοινέ επιλογές προγραμμάτων μέσα στον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για την εργασία σας και τον ενθουσιασμό και να σας ευχαριστήσω διότι ήρθατε ενώπιόν μας και μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς λειτουργεί το ΕΣΕ. Και μέσα στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου θα θέλαμε μεγαλύτερες λεπτομέρειες, διότι θα πρέπει να σας πω ότι με την παρουσία σας αυτή θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές τι πρέπει να διορθώσουμε, ξεκινώντας με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο ένα από τα σημαντικότερα σημεία που θα πρέπει να αποφασίσουμε για το εγγύς μέλλον είναι κατά πόσο είναι κατάλληλη η διάρθρωση του ΕΣΕ ή θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι και να περάσουμε σε μία διάρθρωση του άρθρου 171 πρώην, τώρα 187. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση, στην έκθεση της ομάδας. Ε, καταρχήν ήταν εξαιρετική η έκθεση, θα πρέπει να πω, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, άλλα πρόθεσμα και άλλα μακροπρόθεσμα. Και ανοίγει η πόρτα για μία νέα διάρθρωση του ΕΣΕ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Εάν σε δύο χρόνια ε, περάσει αυτή η απόφαση, δυνάμει του άρθρου 187, κατά πόσο διενεργούνται έρευνες, υπάρχουν ομάδες εργασίας, γιατί θα πρέπει να προβάλλουμε εναλλακτικές, έτσι ώστε να ξεκινήσει το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον ε, πρόεδρο, τον κύριο Μετέη, κατά πόσο η, Επιτροπή σκέφτεται κάτι τέτοιο και τον κύριο Μέννη να τον ρωτήσω τι επιχειρήματα υπάρχουν υπέρ του άρθρου 187 για να περάσουμε στο άρθρο 187. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για το δημοσιονομικό πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό που προβλέπεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για τα 7 χρόνια, θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπετε μέχρι το 2013 γιατί δεν δίνονται πια τόσες υποτροφίες σε εξαιρετικά προγράμματα γιατί δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Και θα ήθελα να σας πω, γιατί και οι, οι τρεις σας είπατε ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη ιστορία, με μια ιστορία μεγάλων επιτυχιών και θα πρέπει να προχωρήσουμε με μια θετική στάση ζωής. και θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα από σας να μου πει τι θα αλλάζετε για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Μερσή λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γκουτιέρες Κορτίνες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα οποία έχουν λάβει η χώρα σε ένα κόσμο θαυμάσιο όπου δεν υπάρχουν προβλήματα με έφεραν οι καλεσμένοι μας. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Η Ευρώπη υποστηρίζει τους ε, ερευνητέ οι οποίοι κάνουν ένα έργο το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι ατομικό, μεμονωμένο. Εγώ όμως πιστεύω ότι με την ε, αντιμετώπιση και την αντίληψη που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, τα κενά που υπάρχουν σε σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχουν πάρα, πολλοί, πάρα πολλές χώρες οι οποίες δίνουν παραγωγικά υποτροφίες για περαιτέρω κατάρτιση στους ερευνητές. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, στις εμπειρίες αυτές που είχατε με πολλούς νέους ερευνητές, μήπως θα ήταν χρήσιμο και ενδιαφέρον να υπάρξει κάποια σύσταση για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς με την Ευρώπη της έρευνας. Πρέπει εμείς να διαχειριστούμε σωστά τα κονδύλια μας και πρέπει να έχουμε και ηγετική στάση σε σχέση με τις βασικές, τα βασικά σημεία εστίασης της έρευνας στο ΜΕΝ. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να αντλήσετε σαν εμπειρία από τους νέους ερευνητέ, πρέπει να τις μεταφράσετε, να μεταφράσετε σε προτάσει. Πρέπει να συλλέξετε την εμπειρία του και να τι μεταφράσετε σε νέε ιδέε. Επιπλέον, θα πρέπει να του δώσουμε δυνατότητα, να, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια αξιολόγηση αναχώρα ώστε να μπορείτε να κάνετε προτάσει σε διάφορε περιπτώσει. Παραδείγματο χάρη στη δική μα περίπτωση τη Ισπανία, όπου σα λέω ότι υπάρχει μια χωριστή, ένα χωριστό φορέας που δίνει τι υποτροφέ από αυτόν που εγκρίνει τα προγράμματα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη ε, συνεκτικότητα μεταξύ προγραμμάτων και χρηματοδότηση με υποτροφίας και έρευνα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα. Αν ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει του σκοπέλου πρέπει να περάσει ένα οποιοδήποτε ερευνητή. Εγώ ήμουνα καθηγητή πανεπιστημίου και βλέπω μεγάλα προβλήματα να βρω ανθρώπους για να έρθουν στο πανεπιστήμιο και να ασχοληθούν με την έρευνα. Γιατί είναι σαν ιεραπόστολος πια ο ερευνητής. Παλιά πήγαινε στην Ινδία σε επικίνδυνες συνθήκες. Κάπως έτσι είναι και οι νέοι ερευνητές σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις δυσκολίες που έχουν μπροστά τους οι ερευνητές. Δεύτερον, εγώ χαίρομαι για την ειλικρινιά σας για το θέμα της ε, γραφειοκρατίας. Και εμείς είμαστε όμοιροι μιας γραφειοκρατίας ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν έχουμε την κάρτα επιβίβασης ή την έχουμε χάσει βγαίνοντας από το αεροπλάνο, δεν μας πληρώνουν δεκάρα. Αυτή είναι λοιπόν μια στάση η οποία είναι μια στάση καχυποψίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για τους ερευνητές λοιπόν δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο λέγεται στο άρθρο 186. Γιατί η γραφειοκρατία είναι ως μια λερναία ύδρα που αποκτά όλο και περισσότερα πλοκάμια. Μεγαλώνει, μεγαλώνει η λερναία ύδρα και τρώει και τρώει όλο και περισσότερου. Επομένω, σα θέτω αυτό το ερώτημα. Πώ θα αντιμετωπίσετε τη γραφειοκρατία. Τρίτο ερώτημα πολύ σημαντικό για μένα. ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά. Τι γίνεται με τι ανθρωπιστικέ επιστήμε. Ποιο είναι ο χώρο ο οποίο αποδίδεται στι ανθρωπιστικέ ε, επιστήμε στον τομέα τη έρευνα, Ποια απάντηση μπορείτε να δώσετε σε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος. Μπορέα Δεκάμπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα. Αυτό το πρόγραμμα έχει πολύ καλή φήμη, όχι επειδή μας είπατε όσα μας είπατε, αλλά γιατί και οι πελάτες σας είναι ευχαριστημένοι από το πρόγραμμά σας. Στην ε, χώρα μου γνωρίζω δύο δικαιούχους του προγράμματος. Επίσης, ε, οι πόροι είναι λογικοί οι πόροι που διατίθενται είναι λογικοί με βάση την ευρωπαϊκή παράδοση. Επίσης βασιζόμαστε στα νέα ταλέντα έτσι ώστε να τους αναθέσουμε τις ανάλογες ευθύνες. Ως προς τα starting grants και τα advanced grants, αυτό είναι κάτι το ιδεώδες διότι μας επιτρέπει να έχουμε μια συνεχή κατάρτιση έχουμε όμως ορισμένες αμφιβολίες. Σε, μια, σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής ασυμμετρίας στον ερευνητικό τομέα. Στα πλαίσια της κινητικότητας των ερευνητών, δεν ξέρω κατά πόσο η κατανομή αναχώρα είναι καλή, διότι εδώ υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κρίσιμη μάζα στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Έτσι ώστε να μην γίνει μία κατανομή υπέρ των πλέον δυνατών. Επίσης υπάρχει ένας κίνδυνος έτσι ώστε ε, ερευνητές, ε, πολύ καλοί ερευνητές να γίνουν μέτροι γραφειοκράτες. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Επίσης, ως προς τα κριτήρια επιτυχίας του προγράμματος, είχαμε 400 δημοσιεύσεις για χίλιες ε, περίπου υποτροφίες. Δεν είναι και εξαιρετικές οι επιδόσεις, αλλά τα κριτήρια επιτυχίας είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων ή θα πρέπει να γίνεται και μία εκ των υστέρων δηλαδή αξιολόγηση. Θα πρέπει να υπάρχει και μία ενδιάμεση αξιολόγηση να περάσουμε από το starting grant στο advanced grant. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση ή πεθαίνουν αυτά τα προγράμματα από φυσικό θάνατο. Για μερικά ισχύει κάτι τέτοιο όπως ισχύει και για το βιολογικό μας κύκλο. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στα πλαίσια αυτού του pipeline θα πρέπει να υπάρχει μία εγγύωση μέσα στα πλαίσια των 150 εκατομμυρίων ετησίως. Ας ελπίσουμε να ισχύσει μέχρι το 2013. Αλλά το θέμα που έχει ως εξής. Από τις διαφάνειές σας είδα ότι υπάρχουν φιλοδοξίες μέσα στα πλαίσια του National Science Foundation, δηλαδή να μετατραπούμε σε, έναν, ένα πλαίσιο ε, εθνικού συνδέσμου. Η National Science Foundation όμως είναι ένας εξαιρετικός ε, οργανισμός. Όμως, πώς μπορούμε να ε, εγγυηθούμε τη χρηματοδότηση πέραν του εβδόμου προγράμματος. Σε πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ματίας, έχετε λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις, τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τις απόψεις και τα σημεία που μας επεσήμεναν. Με προλάβανε οι συνάδελφοι και χωρίς καμιά ντροπή μου κλέψαν τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω, αλλά εγώ θέλω να θέσω ακόμα ένα-δύο ερώτηματα. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία που επέχει η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του για την κυρία Νοβότνη, θα ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει το Mode 1 και το μετά το Mode 2 σε ό,τι αφορά την παραγωγή, την πληροφορία γνώσης. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας είναι πράγματι σημαντικό να υπάρξει αυτή η αλλαγή που αναφέρετε. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία διαιωνίζονται αυτά που είπε ο προλαλής σας για το σύστημα χρηματοδότησης και σχεδιοποίησης. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την προαναφερθήσα απλοποίηση. Πώς λοιπόν λειτουργεί αυτή η διαδικασία της απλοποίησης στο σύστημά σας. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί απόλυτα το επιστημονικό με το, με το γραφειοκρατικό πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα για να επιτευχθεί αυτή η απλοποίηση τα συστήματα υποτροφιών και χορηγήσεων μπορεί να είναι ένας καλός μηχανισμός, αλλά πολλές φορές θέτω αυτό το ερώτημα, γιατί πρέπει τελικά να μιμούμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουμε τα ίδια πράγματα στα οποία εμείς ερχόμαστε πάντα δεύτεροι και καθυστερούμε. Το βασικό μου ερώτημα και κλείνω εδώ είναι είναι το κατά πόσο μπορεί να είναι ένας παράγων αλλαγής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας γιατί τίθενται προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά εδώ και ένα από αυτά είναι το θέμα της συγκέντρωσης των πόρων. Εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα αυτό σημαντικό το ότι πρέπει να συγκεντρώνονται οι πόροι για να γίνεται... Πώς μπορείτε λοιπόν να εξασφαλίσετε ότι θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, γιατί έχουμε τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μερών με τους ερευνητικούς τομείς που έχουν Αυτές λοιπόν οι διαφορετικέ διαφορές που υπάρχουν μέσα στα κράτη-μέλη και μεταξύ κρατών μελών μπορούν να είναι τροχοπέδες για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην Ευρώπη και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως συντελεστής αλλαγής στον ερευνητικό χώρο αλλά δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε και εδώ μεταφέρω κάτι το οποίο το έχουν πει και πολλοί άλλοι, εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο της κυρίας Νοβότνη, για να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος ότι θα πρέπει, συγκεκριμένα όπως είπε η κυρία Νοβότνη, ότι η γνώση πρέπει να είναι και κοινωνικά χρήσιμη η γνώση και αυτό δεν αφορά μοναχά την Ευρώπη, αφορά όλο τον ε, παγκόσμιο χώρο και νομίζω ότι το Συμβούλιο σας μπορεί να συμβάλλει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Äh, Ευχαριστώ. Η κυρία Κολάσκα Μπαμπέντσκα, τελευταία μιλήτρια. poszczególnych krajach Unii Europejskiej, poszczególne kraje Unii Europejskiej bardzo... Εάν ε, δούμε τις ε, διάφορες ε, χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ότι χρησιμοποιούν τα, τους διαθέσιμους πόρους κατά διαφορετικό τρόπο. Μπορείτε να μας απαντήσετε γιατί υπάρχουν αυτές οι, οι διαφορές. Ε, λαμβάνω υπόψη ιδιαίτερα τις χώρες που έχουν πρόσφατα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βρίσκονται πιο πίσω από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι νομίζετε ότι βρίσκεται πίσω από αυτό. Νομίζω ότι οι διαφορές αυτές ένα και θα επιταθούν εάν συνεχίσουμε να προβάλλουμε την καινοτομία, που είναι βέβαια κάτι το φυσικό και πρέπει να το προωθήσουμε, αλλά εάν υπάρχει τεχνολογική ανάπτυξη, οι χώρες που βρίσκονται πίσω θα εξακολουθήσουν να χωλένουν όσο περνάει ο χρόνος, ιδιαίτερα εάν ε, θέσουμε την καινοτομία ως κάτι το πρωταρχικό. Ευχαριστώ. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τον χρόνο μας, αλλά τουλάχιστον υποβάλλαμε όλες τις ερωτήσεις που υπήρχαν. Τώρα θα ρωτήσω τους κυρίους και κυρία εδώ να είναι αναλυτική μεν σύντομοι δε στις τους. Ο καθένα ίσω θα απαντήσει ένα τμήμα των ερωτήσεων. Η καθηγήτρια κυρία Νεβάτα έχει το λόγο. Ναι, θα αξίσω εγώ. Να σας πω ε, για την επιτυχία, πώς βλέπουμε την επιτυχία του ΕΣΕ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το, το φιλοσοφικό υπόβαθρο του ΕΣΕ. Δηλαδή βασίζεται σε ε, μεμονωμένους ερευνητές και μία προσέγγιση bottom-up. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη την δυναμική πορεία της ε, επιστήμης, διότι βρισκόμαστε κοντά στις ενδιαφέρουσες ιδέες και πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτούς τους επιστήμονες. Ιδιαίτερα για την επόμενη γενεά των ε, Ευρωπαίων ερευνητών για να παραμείνουν στην Ευρώπη ή να επιστρέψουν αν βρίσκονται εντός και να είμαστε και δελεαστικοί για τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, το ΕΣΕ λειτουργεί ως παράδειγμα ορίζοντας προδιαγραφές. Οι αξιολογήσεις δεν είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και οι νέοι ε, έχουν άποψη περί δικαιότητας, δικαιοσύνης, με συγχωρείτε, και διαφάνειας του συστήματος ξέρουν εάν έτυχαν ε, δίκαιης μεταχείρισης ή όχι. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έφνης δύο χώρες ε, οι, οποίοι, οι οποίες δεν έχουν την ίδια διαδικασία αξιολόγησης και οι νέοι ζητούν να γίνει αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτή την περίπτωση. Εμείς αποτελούμε ένα λαμπρό παράδειγμα και εδώ θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη διοικητική ευελιξία και μεγαλύτερη καινοτομία μέσα στα πλαίσια το, της προϋπάρχουσας εργασίας, δηλαδή να απλουστεύσουμε ε, μία διοικητική πλαισίωση. Έχετε τα αριθμητικά στοιχεία και μπορείτε να τα συμβουλευτείτε. Θα ήθελα να επανέλθω στις ε, ανθρωπιστικές ε, μελέτες και τις ε, κοινωνικές επιστήμες πάντα είχαν πολύ καλή θέση στο ΕΣΕ και δεν ετέθηκαν το ζήτημα αν ανήκουν εκεί ή όχι. Ανήκουν βεβαίως. Το 14% μάλλον το 10% αφορά ε, όλους τους τομείς και έχουμε ένα επιπρόσθετο 14%. Είδαμε λοιπόν ότι τα αριθμητικά στοιχεία για τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές αυξάνονται, διότι πρόκειται για δύο κοινότητες που ανακαλύπτουν ότι το ΕΣΕ ε, κινείται και προς, αυτούς, προς αυτές τις επιστήμες μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης ε, bottom-up. Και ως προς τη συγκέντρωση πόρων και το, την ασύμετρη κατανομή που υπάρχει, Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να αποτελέσουμε ε, παράδειγμα, διότι η χώρα που μας ρώτησε γιατί, υπάρχει, γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές σχετίζονται με τις χώρες που δεν ε, επενδύουν αρκετά στην έρευνα και στην εκπαίδευση και υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ των επενδύσεων στη χώρα και των, ε, των βοηθημάτων και των ε, χορηγήσεων από το ΕΣΕ. Γιατί δεν διαθέτεται συγκεκριμένα ποσά, ποσοστιαίες αναλογίες, 1-2-3% των διαρθρωτικών ταμείων που να κινηθούν προς, τις ε, βασικές, προς τη βασική έρευνα στα διαρθρωτικά ταμεία αυτό, έτσι ώστε να φτάσετε σε επίπεδο, στο επίπεδο να μπορέσετε να ανταγωνιστείτε ε, και στο ΕΣΕ. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα ενθαρρυντικά μηνύματα. Στο Βουκουρέστι συζητήσαμε με τους ε, Ρουμάνους συναδέλφους και το βασικό μήνυμα είναι να υπάρχουν αρχές αριστείας στην ίδια τη χώρα, να μην γίνονται παραχωρήσεις και υποχωρήσεις και έτσι ενισχύονται αυτές οι χώρες. Αλλά και οι χώρες αυτές θα πρέπει από τη δική τους πλευρά να δημιουργήσουν τους απαράβατους όρους στα ε, πανεπιστήμια τους όπως γίνεται τώρα στην, Πολωνία έτσι ώστε να αρθεί στο, στο ύψος των, των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ευχαριστώ. θα αρχίσω από το σημείο στο οποίο εσείς ε, τελειώσατε. Σίγουρα θα περάσει χρόνος μέχρι ότου τα, τα νέα κράτη-μέλη προλάβουν τα προπορευόμενα παλιά κρατημέλη στα θέματα της έρευνας. Πρώτα απ' όλα όμως, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίς. Παραδείγματος χάρη, βάσει της ε, προηγούμενης μου εμπειρίας, είχαμε πάρα πολλούς, ε, ιδιαίτερα λαμπρούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές για διδακτορικό, από την πολιτεία. Βέβαια θα χρειαστούν πολλά χρόνια αυτοί να γίνουν ακαδημαϊκοί, οι οποίοι θα μπορούν να συναγωνίζονται με αυτούς από τα παλιά αλλά δεν πρέπει να προσπαθήσουμε με ένα τεχνητό τρόπο να εξισώσουμε όλους αυτούς τους φοιτητές. Ή θα πρέπει να γίνουμε Κινέζοι. Οι Κινέζοι στέλνουν τους φοιτητές τους παντού, σε όλο τον κόσμο, Δύο Συνομές Πολιτείες για να έχουν την καλύτερη εκπαίδευση και μετά τους επαναπατρίζουν τους καλύτερους φοιτητές τους από όλε τι χώρε του κόσμου. Και αυτή η κινέζικη στρατηγική απεδείχθη πάρα πολύ χρήσιμη και ταχεία. Ένα τρόπο είναι αυτό. Ένα άλλο τρόπο, ο οποίο μπορεί να μα οδηγήσει επέκεινα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα, έχει να κάνει με την χρηματοδότηση με τις υποτροφίες Μαρία Κιουρί. Θα μπορούσαν να διευρυνθούν αυτέ οι υποτροφίες. Γιατί αυτές οι υποτροφίες είναι ένα είδος μεταδιδακτορικού ε, μεταδιδακτορικής υποτροφίας ή χορήγησης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια έλλειψη τέτοιων χορηγήσεων υποτροφιών για τους μεταδιδακτορικούς επιστήμονες. Υπάρχουν περίπου 60.000 τέτοιες υποτροφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο τρίτα αυτών δίδονται σε μη Αμερικανούς. Και η επιτυχία της Αμερικανικής έρευνας είναι ότι μπορεί να είναι τόσο ελκυστική για νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης, ο οποίος είναι ο ηγέτης μιας ε, ε ιδιαίτερα φημισμένης ερευνητικής ομάδας σε ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα μόνο 10% των ερευνητών στην ομάδα αυτή των, των συνεργατών του θα είναι Αμερικανοί. Γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει καταρχήν να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ στο να κρατήσει όσο πολύ, όσο περισσότερους μεταδιδακτορικούς υποτρόφους στην Ευρώπη ή να καταφέρει να τους επαναπατρίσει ή να προσελκύσει τους Κινέζους, τους Ινδούς και τους άλλους στην Ευρώπη, ώστε να ενισχύσει τις ερευνητικέ ομάδες στην Ευρώπη. Μπορώ να σας πω, αυτό είναι μια προσωπική, αν θέλετε, υπενθύμηση. Εγώ έχω εκπαιδευτεί σε ένα γαλλικό ε, επαρχιακό πανεπιστήμιο. Και όταν πήγα στη συνέχεια Ηνωμένε ΗΠΑ ω μεταδιδακτορικός ερευνητής, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και ήταν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου. Έμαθα τι σημαίνει πραγματική βιβλιοθήκη, παραδείγματο χάρη, και πολλά άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε λοιπόν πολύ περισσότερε ευκαιρίε στου καλύτερου επιδικατορία φοιτητέ μα και στου αντίστοιχου από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θα πρέπει να χρειάζονται έξι μήνε από τη στιγμή που δίδεται μια υποτροφία Marie Curie και το χρόνο που τελικά ξέρει αυτός που πήρε την υποτροφία πόσα λεφτά θα πάρει. Έξι λεφτά είναι. Έξι μήνες είναι πάρα πολύ για να υπάρξει η τελική σύμβαση όταν αυτό είναι απαραίτητο. Είναι σημαντικός ο χρόνος αυτός. Μπορούμε να απλοποιήσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή διαχείριση, η χρηστή διαχείριση, να είμαστε υπόλογοι κτλ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν φταίμε εμεί για όλα αυτά που έχουν γίνει με την Επιτροπή Σαντέρ πριν από 15 χρόνια. Μετά από το, την εποχή αυτή όλοι έχουν γίνει καχύποπτοι. Α το ξεχάσουμε αυτό, ας φτιάξουμε μια συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει απάτες θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιε και αυστηρέ κυρώσει. Αλλά δεν μπορείτε τώρα να έχετε μία επιτροπή που απαρτίζεται από εξέχοντες επιστήμονες να ελέγχουν τα, τις κάρτες επιβίβασης και τα εισιτήρια τρένων. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτά που είναι σημαντικά και όχι σε αυτά τα οποία είναι δευτερεύοντα. Χρηματοδότηση. Είναι σημαντική η χρηματοδότηση. Δεν είναι όμως ο αποφασιστικός παράγων. Αν δεν υπάρχει καλή διαχείριση της χρηματοδότησης, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Κάποιοι οι οποίοι χρειάζονται περισσότερα λεφτά, εντάξει πρέπει να διορθωθεί αυτό να έχουν περισσότερα λεφτά στο μέλλον. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο, ο φορέα, ο χρηματοδοτικό να έχει την αυτονομία και την ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά τα πόσα αυτά. Δεν είναι το σημαντικό να δώσετε περισσότερα λεφτά στο φορέα μα. Και η κινητικότητα των επιστήμων είναι πολύ σημαντική αλλά και η κινητικότητα μπορεί να ευνοηθεί με άλλα μέσα, όπως παραδείγματος χάρη υποτροφίες Marie Curie. Υπήρξε επίσης ένα ερώτημα για το αν θα πρέπει να μεταμορφώσουμε, αν πρέπει να, αν αυτό που κάνουμε μεταμορφώνει τους νέους ερευνητές σε εμπειρογνώμονες στη διοικητική διαχείριση. Είναι γεγονό. Σε πολλέ χώρε, όπω και η δική μου, πολλά πανεπιστήμια δεν μπορούν να κάνουν αιτήσει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν δημιουργήσει ειδικέ μονάδε για να μπορούν να συμπληρώνουν τι αιτήσει. Δεν μιλάω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνε. Μιλάω για άλλα προγράμματα μέσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αν σε μια γραφειοκρατική χώρα σαν τη Γαλλία, με γραφειοκρατική παράδοση, θέλετε να έχετε ειδική εμπειρογνωμοσύνη για να υποβάλλετε προτάσεις, Κάτι δεν πάει καλά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια απλοποίηση ιδίω του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό είναι προαπαιτούμενο αν θέλετε πραγματικά να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια με έναν τρόπο που είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα να ευχαριστήσω την κυρία Καβάρη για την ερώτησή σα, γιατί μου κάτι Το ε, τ είναι μια που, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σύγκριση. Το είχε εμπνευστεί από το ΕΣΕ στο παρελθόν. Μετά είχαμε κάποιε δυσκολίε. Σήμερα θα πρέπει εμείς να εμπνευστούμε από το ΙΑΙΤ. E το πρώτο είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιότυπο σχέδιο, εν αντιθέσει προς το ΕΣΕ. Ίσως αυτό είναι εξής πραγματικά το σκεφτούμε. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά γιατί εδώ έχουμε μια ε, συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και η έρευνα εχνής είναι πάρα πολύ θέμα του δημοσίου τομέα. Απλούστευση. Φυσικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Έχουμε τώρα κάποιες ε, χορηγήσεις σε απλουστευμένα προγράμματα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμη πιο απλουστευμένο και να χορηγούνται ε, κάποιες ε, χορηγήσεις ε, διαφορετικά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και από την άλλη μεριά ενδιαφερόμαστε να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις για την αναθεώρηση των διαδικασιών. Αυτά βέβαια είναι θέματα δημοσιονομικά. Τα συστήματα αξιολόγησης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως είπε και η Χέλγα προηγουμένως. Ορισμένε χώρε λένε σα παρακαλώ βοηθήστε με για να διατηρήσουμε αυτή την έννοια τη ε, αριστεία. Και η περίπτωση τη Ρουμανία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί όταν συζητήσαμε με τον ε, Ρουμάνο Υπουργό, νέο επιστήμονα, είπε ότι πραγματικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητε. Έχουν καταπληκτικά πράγματα να προσφέρουν και ένα τμήμα των ε, Ρουμανικών διευθυντικών ταμείων θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιηθούν ε, μέσα σε πλαίσια πλασφόρμα CNC για ε, e για, τους, για τα κέντρα αυτά αριστείας. Τώρα, για το προπολογισμό, 7,9 δις ευρώ ήταν καλό κεφάλι να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά πτυχές 12-15% είναι πάρα πολύ σωστά. Πραγματικά εμείς είμαστε top. Αυτό το βέβαια είναι σωστό. Αυξάνεται ο όγκος των αιτήσεων και οπωσδήποτε θα έχουμε νέα μέσα που θα προωθηθούν και θα θέλουμε περισσότερους πόρους στο μέλλον. Έχουμε ένα πολύ καλό σημείο κίνησης το σημείο συνάντησης είναι σε δύο χρόνια, ε, το 2011 δηλαδή, και μπορώ να σας πω ότι η νέα επίτροπος κυρία Γκέγκαν είναι πάρα πολύ δεσμευμένη να πετύχει αποτελέσματα. Εργάστε πάρα πολύ σοβαρά επισκέφθηκε το Συμβούλιο, συνάντησε την Χέλγκα Πραγματικά έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα από αυτή τη πλευρά. Είναι μια πρόκληση για μας. Για τις περισσότερες συστάσεις θα έλεγα. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε σημαντική πρόοδο. Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού βέβαια είναι ακόμα ένα ανοιχτό ερωτηματικό. Τι θα άλλαζα. το πρότυπο των ε, ε, χορηγήσεων και υποτροφιών και επίσης το θέμα των ελέγχων δεν μπορούμε να έχουμε τε, καθημερινό έλεγχο από την αρμόδια γενική διεύθυνση γιατί αυτό δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης. Τώρα, κατά πόσο οι κύριοι ερευνητέ ε, μετατρέπονται σε γραφειοκράτε, όπως είπε ο κ. Κοριαντεκάμπος, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και εγώ είχα την εκπαίδευσή μου στις ΕΙΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της ε, Καλιφόρνια, που είναι από τα καλύτερα. Και εκεί υπήρχε μια πτυχή διαχείρισης. Πάντα χρειάζεται διαχείριση όταν κανένας έχει στα χέρια του ε, δημόσια χρήματα. Η αμερικανική πλευρά όμω μπορεί πολύ αποτελεσματικά να αφαιρέσει το της εργαφραγητές από τους ερευνητές και να το αναλάβει το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο. Εμείς πραγματικά έχουμε πολύ καλούς ερευνητές στο ΕΣΕ και μας έχει εντυπωσιώσει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται. Βρισκόμαστε στη Ρωστή Άγουσα. Κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε εμείς ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκού τύπου ε, Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σαν το NSF. Διαφέρει η Ευρώπη βέβαια από τη ΣΥΠΑ. Τώρα νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ. Απάντησα στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ καθηγήτρια κυρία ε, Νοβότμη, κύριε Μένη, κύριε Μέτρη, νομίζω ότι ήταν ε, πραγματικά μια καλή διαφήμιση στην ευρωπαϊκή πολιτική έρευνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ό,τι καλό στο μέλλον, καλή συνεργασία με εμά και επίσης να διατηρήσετε την απαραίτητη ανεξαρτησία που είναι απαραίτητη. Και αν χρειαζόστε τη βοήθειά μας, να έρθετε εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ε, ολοκληρώνουμε με αυτέ τι μεσαίε και περνάμε στο επόμενο. Merci. Meine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 Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Προσπαθώντας το σύντομο του χρόνου που έχουμε, να εξετάσουμε το τόσο σημαντικό αυτό σημείο. Είχαμε αναθέσει μια μελέτη για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροφαγική βιομηχανία. Έχουμε τα αποτελέσματα εδώ. Θα ακούσουμε κάτι σχετικά χαιρετίζω την Άννα Σοφία Κέρσου Ζαμπράκο και τον Φερνάντες Πένα. Δεν ξέρω αν τα πρόφερα σωστά τα ονόματα. Σας χαιρετίζω πάντως. Μπορείτε να αρχίσετε. Μόλις αρχίσει το μηχάνημα λειτουργεί. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης σε σχέση με τις συνέργειες μεταξύ του αυτοκινηστικού και του αεροναυτικού τομέα και της αλυσίδας προμηθευτών τους. Η μελέτη αυτή έγινε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου το 2008 και το 2009. Πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Επομένως πρέπει να τα δείτε αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, θα ξεκινήσω με την παρουσίαση τις εταιρείε που ήταν υπεύθυνη για αυτή τη μελέτη, τη ΣΥΝΤΟ, είναι ένα κέντρο στην Ισπανία για την έρευνα στην ενέργεια και την ανάπτυξη και μετά θα κάνουμε μια παρουσίαση της μεθοδολογίας. και θα δούμε μετά ποια είναι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που μπορούμε να διατυπώσουμε. Εντάξει. Επειδή κάναμε τη μελέτη στα αγγλικά δεν μπορώ να... Είναι πιο εύκολο την παρουσιάσω στα αγγλικά. <laughs> Okay. Bueno, yo voy a... Εντάξει, θα μιλήσω ισπανικά. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Νομίζω ότι λύσαμε τα προβλήματα πληροφορικής και μπορούμε να πούμε ορισμένα σχόλια για τον φορέα από τον οποίο προερχόμαστε και ο οποίος μας επέτρεψε να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνουμε αυτή την έρευνα. Λοιπόν, επομένως, ίσως και χωρίς τις διαφάνειες μπορούμε να προχωρήσουμε. Είμαστε ένα κέντρο μελετών. Ξεκινήσαμε τις ε, έρευνές μας σε ό,τι αφορά τα, τον αεροναυτικό τομέα και τα αυτοκίνητα, αλλά περάσαμε μετά και στον τομέα της ενέργειας και αυτό μας οδήγησε η ίδια η έρευνά μας. Γιατί όλο και περισσότερο βλέπαμε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων και επίσης να υπάρξει μεταλαμπάδευση τεχνολογίας από, την, από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στον αεροναυτικό τομέα, είτε και τούμπαλιν, ακόμα και προς τον τομέα των συντηροδρόμων. Και όλα αυτά είναι δυνατά γιατί, γιατί ένα τμήμα της έρευνας βασίστηκε στην ε, αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για να υπάρξει αυτή η σύνδεση των αναγκών με το τελικό προϊόν. Έχουμε λοιπόν τη γνώση αυτή ως ε, μεμονωμένα άτομα και ως ομάδα για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις αλυσίδες προστιθέμενης αξίες στους τομείς αυτούς. Στον τομέα τον αυτοκινηστικό υπάρχει μεγάλη απέτηση σε ό,τι αφορά τον χρόνο κατασκευής, σε ό,τι αφορά την συμπίεση του κόστους και σε ό,τι αφορά την μεγαλύτερη χρήση τεχνολογίας. Μπορούμε να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, σαν παράδειγμα, Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι, οι εσωτερικές αλυσίδες παραγωγής, μέσω μιας προσωμείωσης μπορούμε να ξεκινήσουμε να περάσουμε σε αρχέτυπα, σε παραγωγή, σε επαλήθευση και παραγωγή σε βιομηχανικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν έχουμε προχωρήσει στη μεταλαμβάνευση τεχνολογίας από ένα φορέα σε ένα άλλο. Νομίζω ότι είναι έτοιμη η παρουσίαση. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να δημιουργήσουμε τα λεγόμενα spin-offs, τις εταιρείες οι οποίες προκύπτουν από τα ερευνητικά αποτελέσματα, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα και φτάνοντας στην εφαρμογή της τεχνολογίας και στον τομέα της αεροναυτικής και στον τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων. Βλέπετε λοιπόν στην ε, διαφάνεια αυτή κάποια παραδείγματα. Τα, η εταιρεία Λεαθιώνες Λιχέρας είναι μια επιχείρηση η οποία παράγει ανταλλακτικά από αλουμίνιο για τα αυτοκίνητα και έχει προχωρήσει σε μια διαργασία που έχουμε σχεδιάσει εμείς πλήρως και τώρα βρίσκεται σε επίπεδο παραγωγής εδώ και μερικούς μήνες και έχουν βγει και τα πρώτα αυτοκίνητα τα οποία παράγονται με αυτή τη διαδικασία και συγχρόνως μπορούν να παράγουν εξαρτήματα για την αεροναυτική βιομηχανία. Πέραμε τώρα στους στόχους της ε, μελέτη και δίνω το λόγο στην Ανασοφία. After this brief introduction, of our Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή θα αρχίσουμε με την βασική μελέτη. Βασικός στόχος είναι να δούμε ποιες είναι οι πολλά υποσχόμενες συνέργειες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε αυτό το συσχετισμό, δηλαδή το, το τομέα των αυτοκινήτων και της αεροναυπηγικής, έτσι ώστε να προτείνουμε συγκεκριμένες συστάσεις για να ενισχύσουμε αυτές τις συνέργειες υπέρ και των δύο τομέων. Έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μελέτη ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Ξεκινήσαμε με ε, μία έρευνα τεκμηρίωσης και μετά προβήκαμε σε μία ανάλυση χρησιμοποιώντας έρευνες και συνεντεύξεις για να ορίσουμε, να ταυτοποιήσουμε αυτές τις συνέργειες και να προβούμε σε συστάσεις. Τα αποτελέσματα ε, ήταν ε, πολύ θετικά, δηλαδή χρησιμοποίησαμε πάνω από 100 έγγραφα Χρησιμοποιήσαμε χαρτογραφήσεις, οδικούς χάρτες και ούτω καθεξής για να μπορέσουμε να προβούμε προς στάσεις. Ο βασικός στόχος είναι να έχουμε μία γνωμοδότηση από τους ε, εμπλεκόμενους φορείς και από τους δύο ε, τομείς υπέρ αυτών των συνεργειών για να μας πούν αν προϋπάρχουν καταρχήν και αν θα ήταν εφικτό να έχουμε κοινοτικέ δράσεις ενίσχυσης. Ήρθαμε σε επαφή με 200 ε, εμπλεκόμενους φορείς από τα πανεπιστήμια, από τη βιομηχανία, καθώς και άλλους φορείς. Και τα βασικά θέματα που ε, ανέκυψαν αφορούσαν αρκετούς τομείς, αλλά αυτό μας ενδιέφερε καταρχήν ήταν οι ενδυνάμεις συνέργειες, εάν υπάρχουν και ανέ, ναι, σε ποιες τεχνολογίες και κατά πόσο θα πρέπει να αναλυφθεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και για τους δύο τομείς και πώς μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Είχαμε ε, στοιχεία από 60 εμπλεκόμενους φορείς, αυτά τα στοιχεία ανάδρασης, καθώς και συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, ε, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, βασικές ευρωπαϊκές ενώσεις, κλέπε, γιόκαρ και άλλους φορείς και περίπου 17 χώρες συμμετείχαν στην διενέργεια αυτής της έρευνας. Ποια ήταν τα αποτελέσματα λοιπόν. Το 80% των εμπλεκόμενων φορέων θεώρησαν ότι υπάρχει αυτή η, δυναμική, αυτό το δυναμικό συνέργειας. Μιλήσαμε για νέα υλικά στα ηλεκτρονικά συστήματα και πάνω το 70% τάχθηκε υπέρ μιας νέας πρωτοβουλίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να προωθηθεί αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ε, Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε σχέση με αυτές τις ε, συνέργειες ε, υψηλών δυνατοτήτων, θα πρέπει να δούμε πώς ισχύουν για τους ε, εμπλεκόμενους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε πώς ένας τομέας μπορεί, μπορεί να ευεργετηθεί από έναν άλλο. Για να ξεπεράσουμε ε, αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να ορίσουμε αυτές τις συνέργειες ως προς το ε, μελλοντικό τους, τις μελλοντικές δυνατότητες, διότι πολλές φορές είναι δύσκολο να τις αναγνωρίσουμε. Οι κύριες τεχνολογίες λοιπόν που έχουν υψηλό δυναμικό για το μέλλον είναι η αλυσίδα προμήθειας, και η διαχείρισή της, πώς μπορούν οι αλυσίδες προμήθειας και των δύο κλάδων να ωφεληθούν από συνέργειες. Μπορεί λοιπόν η κάθε πλευρά να υποφεληθεί από τη συσσωρευμένη εμπειρία της άλλης πλευράς και τούμπλεν. Επίσης, πολλά συστήματα, πολλά κέρια συστήματα που χρησιμοποιούνται στα, στην παραγωγή αυτοκινήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα αεροπλάνα. Αυτό κάνουν ήδη κάποιες πρωτοβουλίες και επίσης η τυποποίηση είναι μια στρατηγική όπου μπορεί να υπάρξει συνέργεια μεταξύ των δύο τομέων. Από τεχνολογική πλευρά. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους περισσότερους εμπλεκομένους είναι τα νέα ε, υλικά τα, οι ανοιχνευτές, οι φωτονικοί, τα ΕΦΗ συστήματα και τα συστήματα πλοήγησης. Αυτά που θεωρούν ότι έχουν υψηλή ή τουλάχιστον μέση δυνατότητα ανάπτυξης και μπορεί να είναι υψηλή δυνατότητα μελλοντικού δυναμικού, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη ακόμα η ανάπτυξή τους, είναι τα θέματα αναλλακτικών καυσίμων και οι δύο τομείς εργάζονται στους τομείς αυτούς αλλά ο τομέας των αυτοκινήτων είναι πολύ πιο προχωρημένος και επειδή είναι διαφορετικές οι απαιτήσει στους δύο τομείς, δεν είναι φανερό πώς μπορεί να μεταλαμβαδευτεί η τεχνολογία από τον ένα τομέα στον άλλο. Επίσης, <clears throat> αυτό συμβαίνει και με την μείωση του θορύβου. Εκεί που υπάρχει μεσαία και υψηλή ικανότητα δυναμικού στο μέλλον, όπου η τεχνολογία είναι με πολλές ελπίδε. αλλά δεν σαφές πώς μπορεί να υποφεληθεί από συνέργειες, είναι η ανακύκλωση. Ο τομέας των αυτοκίνητων, όπω γνωρίζουμε πολύ καλά, έχει αυστηρού κανόνες για την ανακύκλωση, κάτι που δεν συμβαίνει στην αεροναυπηγική, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο και υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη που εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή βιομηχανικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες από την Airbus και την Boeing. Είναι ένα τομέα λοιπόν που θα είναι ενδιαφέρον να έχουμε περαιτέρω συνεργίες στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Εκεί που είναι χαμηλότερη η δυνατότητα για το μέλλον ή που ο αντίκτυπος ο δυνητικός τους δεν είναι τόσο σημαντικός αυτών των συνεργειών, είναι η δοκιμασία συστημάτων, ίσως για τα ελικόπτερα και τα μικρά αεροσκάφη, γιατί για τα μεγάλα αεροσκάφη δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρξει κοινή δράση στους, στον τομέα της δοκιμασίας. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίε εκεί, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο δυναμικό εκμετάλλευσης με χαμηλό δυναμικό. Έχετε το θέμα των κινητήρων, συστημάτων τροχοπαίδησης, αλλά και υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει στις δύο περιπτώσεις και δεν μπορούν να μεταφερθούν παραγωγός χάρη οι μηχανές από τα αεροσκάφη στα αυτοκίνητα. Κάποια μικρά αεροσκάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτο, μηχανές αυτοκινήτων. Είναι κάποιε πρωτοβουλίε οι οποίες όμως δεν έχουν καρποφόρηση ακόμα. Επίσης για τα συστήματα ε, τροχοπέδησης, τα συστήματα όρασης υπάρχει κάποια κοινή δράση. Επομένως, επί τη βάση όλων αυτών και επί τη βάση των πρωτοβουλειών που έχουμε μελετήσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες δράσεις, καταρχήν για να προωθήσουμε συνέργειες σε βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι σαφείς οι συνέργειες και σε άλλες περιπτώσεις είναι η συνέργεια. Αλλά είναι ασαφές το τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση αυτών των συνεργειών. Για τις βραχυπρόθεσμες δράσεις, οι εμπλεκόμενοι πιστεύουν ότι τα υπάρχοντα εργαλεία, όπως είναι το πρόγραμμα πλαίσιο 7 για την ε, έρευνα, μπορούν να προωθήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα νέα υλικά, με τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα πληροφορικής, πλοήγησης και την ανακύκλωση. Πολλά πρέπει να γίνουν επίσης σε σχέση με τα πρότυπα, σε συνεργασία με τη ΣΕΝ, επί τη βάση του, της που γίνεται από τον τομέα αυτοκίνητο βιομηχανίας. <clears throat> Μπορούν επίσης πολλά να γίνουν μέσα στην ΣΥΠ, να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη μεταλαμπάδευση γνώσης με, σε σχέση με τις αλυσίδες προμήθειας. Για τις μεσοπρόθεσμες δράσεις, αυτές είναι δράσεις που δεν αφορούν νέα προγράμματα κυρίως, αλλά που αφορούν να υπάρχει καλύτερη έρευνα στο να ξέρουμε τι μπορεί να μεταλαμπαδευτεί από τον ένα τομέα στον άλλον. Εναλλακτικά καύσιμα, όπως είπαμε και όπως εξήγησα προηγουμένως ενδελεχώς. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών πλατφορμών που εργάζονται στα θέματα αυτά, όλες από τις οποίες έχουν μια πληθώρα εγγράφων σε σχέση με τα θέματα αυτά. Και όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους, εάν συνεργαστούν και προσπαθήσουν να δουν τι μπορούν να κάνουν μαζί. επομένω. Έχουμε ενώπιον μας μια ευκαιρία να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την έρευνα η οποία γίνεται και για τους δύο αν συνεργαστούν. Και με τον τρόπο αυτό να έχουμε μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα. Έχουμε οκτώ συστάσεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει για να εξασφαλίσουν την πρόθεση αυτών των συνεργειών που θα επιτρέψουν να μειωθεί και το κόστος της έρευνας στους διάφορους τομείς. Παραδείγματος χάρη για τα ενσωματωμένα συστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και στους δύο τομείς. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ώστε να μην έχει ο ένας τομέας διαφορετικά συστήματα ενσωματωμένα από ότι ο άλλος. Οι συστάσει μας λοιπόν τονίζουν ότι είναι καλύτερο να υπάρχει και συντονισμένη, συντονισμός στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν περισσότερες προσκλήσεις για οριζόντιες δράσεις μέσα στον τομέα των μεταφορών για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων που αφορούν το θέμα της αεροναυτικής και της ε, αηφόρου μεταφοράς στο συγχεσαίο επίπεδο μεταξύ των ενσωματωμένων συστημάτων και άλλων υποκατηγοριών. Και όχι μονάχα τα θέματα έρευνας, αλλά και τα θέματα που άπτονται της παραγωγής. Όπως σας είπα, μέσα στο πρόγραμμα συντοώ το θέμα της αλυσίδας προμήθειας για τις, τους δύο τομείς Εξόχως σημαντικό και για τις δύο πλατφόρμες θα είναι όταν καθορίζουν την ερευνητική τους ατζέντα να δουν ποιοι είναι τομείς όπου μπορούν και οι δύο φορείς, οι δύο τομείς να εργαστούν από κοινού και να προτείνουν στην Κομισιόν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αμοιβαίας επωφέλειας Για να μπορέσουν να προωθηθούν τα θέματα αυτά θα είναι επίσης να προωθήσουμε την πρωτοβουλία, τις πρωτοβουλίες εργασίας μεταξύ των ερευνικών συμπλεγμάτων που θα έχει αποτελέσματα θετικά και για τις δύο πλευρές. Και θα είναι επίση ενδιαφέρον να δούμε πώς με χρόνια και καιρούς αυτή η συνεργασία θα εξελιχθεί περισσότερο και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε λοιπόν μια ε, δυνατότητα αξιολόγησης αυτής της συνεργασίας μεταξύ του αυτοκινηστικού και του αεροναυπηγικού τομέα. Και να έχουμε φυσικά και συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Ένα περαιτέρω θέμα το οποίο ανέφεραν σήμερα ορισμένοι ομιλητέ. Είναι ότι αν υπάρχουν κοινέ δράσεις και για τους δύο τομεί. θα πρέπει να γίνεται από κοινού και για τους δύο Τελικές παρατηρήσεις. Κάτι το πιο σημαντικό είναι ότι για οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία να εμπλέκονται και οι δύο τομείς. για να εξασφαλίσουμε ότι το τελικό προϊόν θα είναι πρόσφορο και για τους δύο τομείς. Και για μια τελική τελική παρατήρηση, το έγγραφο αυτό έχει παραχθεί σε ένα αενάως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. Και κάποια από αυτά τα στοιχεία και κάποιες από αυτές τις πληροφορίες έχουν ε, περάσει και μια διαδικασία περαιτέρω εξέλιξης πες, οπότε μπορούμε εν καιρό να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Προσπάθησα να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ και τις δύο ε, κυρίες για την παρουσίαση της μελέτης αυτής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας τα παρουσιάσετε τόσο αναλυτικά. Ε, είναι αρκετό σκορός από τότε που αναθέσαμε τη μελέτη αυτή και δεν μπορούσα να παρουσιαστεί έγκαιρα. Συνάδελφος ο Ντί έχει πρώτο ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ντί. Πάρα πολύ σύντομα πρόεδρε. Η οργάνωσή σας, που είναι μια είναι κυβερνητική οργάνωση, ανήκει σε ποιον. Ποιος επιδρά δηλαδή στην οργάνωση αυτή. Και υπάρχει στην διάταξη, κύριε Πρόεδρε, γιατί εμεί συνανθέσαμε εμεί τη χρηματοδότηση Πώ έφτασε το θέμα αυτό στην ημερήσια μα διάταξη, ίσω κάτι μου έχει διαφύγει. Επίσης αναφερθήκατε στην εξέλιξη των, του αυτοκινητού ε, της αλλά και του σιδηροδρομικού τομέα. Γιατί έχει αστιαστεί η μελέτη αυτή στην βιομηχανία και την ναυπηγική βιομηχανία θα είναι τμήμα μιας συμπληρωματικής ανάλυσης και ο συνδρομικός τομέας. μια πολύ γενική παρουσίαση. Ε, νομίζω θα επανέλθουμε στην Επιτροπή μας κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή για ένα βουλευτή και για ένα πολίτη το ίδιο θα ισχύει. Ένα ερευνητικό κέντρο. Όταν βλέπουμε τι ακούμε για την πολιτική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη-μέλη, καταλήγουμε σε ένα πολύπλοκο δομών, ιδρυμάτων, ε, οργάνω που ασχολούνται με τα πάντα. Κάποια στιγμή θα έχουμε Περθεί τελεία. Ε, ξέρετε ότι συζητάμε για την γεωργία και την έρευνα και λέμε πολλά, θα πανούμε για τη γεωργία, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για την έρευνα, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο είναι αποτελεσματικά οικονομικά τα χρήματα που χρησιμοποιούμε για την έρευνα. Με συγχωρείτε για αυτό το συμπέρασμα που είναι ίσως εκτός θέματος, αλλά ε, δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό σας το παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε, παρακαλώ. Βεβαίως. Ίσως Κάποια από τα ερωτήματά σας αναφέρονται βέβαια στον πρόεδρο της Επιτροπής σας, αλλά αυτά που έχουν να κάνουν με τη μελέτη και την οργάνωση, μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Ρωτήσατε τι φορέας είμαστε. Είμαστε μη κερδοσκοπικό φορέας που κάνουμε έρευνα και είμαστε απόλυτα ανεξάρτητοι. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα άλλο φορέα, ούτε υποκείμεθα στην έλεγχο κάποιου άλλου. Βέβαια, έχουμε τον έλεγχο των κυβερνητικών φορέων και όλα αυτά τα οποία κάνουμε γίνονται για κοινοφελείς σκοπούς. Για το επόμενο ερώτημα που θέσατε, γιατί δεν μιλήσαμε για τον σιδηρόδρομο, συμφωνούμε ότι είναι ένας άλλος νευραλικός τομέας, ιδίως σε σχέση με ορισμένα θέματα, μπορεί να υπάρξει μια μεταλαμβάνευση τεχνολογίας μεταξύ αεροπλάνου, σιδηροδρόμου και αυτοκινήτου. Αυτή τη στιγμή το αντικείμενο της έρευνας περιλάμβανε μονάχα αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Συγκεκριμένα το... η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Κομισιόν περιλάμβανε μονάχα αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όλο και περισσότερο υπάρχουν περισσότερες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να ε, μεταφερθούν από τον ένα των τριών τομέων που αναφέρατε στους άλλους. Και τέλος νομίζω ότι το τελευταίο σας ερώτημα ήταν, εάν δεν με απατάει η μνήμη μας, για τους διάφορους <clears throat> φορείς και τις σχέσεις που έχουμε με αυτούς. Δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο άτομο για να απαντήσω αυτό. Μπορώ να πω είναι ότι αυτή η μελέτη είναι ένα πρώτο βήμα για να εξασφαλίσουμε την ορθολογικοποίηση των δαπανών στους τομείς αυτούς, γιατί δημιουργούνται πολλές τομές, η Ευρωπαϊκή πολιτική όλο και περισσότερο έχει σαν στόχο να μην υπάρξει επικάλυψη ερευνών, να μην γίνονται εργασίες σε διαφορετικές χώρες οι οποίες έχουν το ίδιο ακριβώς αντικείμενο και τον ίδιο στόχο. Μέσα στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι η μελέτη μας προσπαθεί να κάνει ένα βήμα ακόμα προς τα εμπρός, όχι λοιπόν να γίνεται μόνο σε τομείς τεχνολογικούς μονομένου η έρευνα, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε την εγκαρσιότητα και την συνέργεια μεταξύ διαφόρων τομέων, όχι μόνο μεταξύ τεχνολογιών, αλλά και μεταξύ τομέων παραγωγή. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ελπίζω ότι έχουμε δώσει μια απάντηση σε αυτά που είπατε. Έχουμε παρακολουθήσει, λοιπόν, αυτά που έχουν γίνει και φυσικά θα συνεχίσουμε να ερευνούμε τι γίνεται μεταξύ αυτοκινητιστικού τομέα, σιδηροδρόμων και αεροναυπηγικής. Κυρία Τροτουμάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήρθα να παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, παρουσίαση αυτή γιατί ζω σε μία περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα και αριστεία στον τομέα των οχημάτων του μέλλοντος. Βεβαίως μας ενδιαφέρει και η αεροναυπηγική γιατί έχουμε εγκαταστάσεις σε αυτή την περιφέρεια της Γαλλίας, της Ανατολικής Γαλλίας και βεβαίως έχουμε και έναν πυρηνικό σταθμό. Υπάρχουν λοιπόν ε, υπάρχουν αυτοί οι σύνδεσμοι ή μεταφοράς δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κρίσης. Αυτό δεν αφορά μόνο τους κατασκευαστές. Εγώ είχα πολλές προσδοκίες από αυτή τη μελέτη. Καταρχήν να δούμε ποιες είναι οι εμπλεκόμενες βιομηχανίες. Είναι οι κατασκευαστές, αυτοί που αναλαμβάνουν ε, υπεργολαβίες, ποιοι από όλους. Έπειτα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σήμερα στην αεροναυπηγική, στην αυτοκινητομηχανία επίσης και στο τομέα των ενεργειακών καυσίμων ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το, και τον τομέα της απασχόλησης έτσι ώστε να βρούμε συγκεκριμένες ε, απαντήσεις. Αυτό αφορά την διαχείριση, τα ΤΕΙΣΕ, την ε, έξυπνη ενέργεια θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα διαχειριστούμε. Όμως θα πρέπει να φτάσουμε σε μία μεθοδολογία από τη μελέτη σας. Εσείς κάνατε κατανομή σε τρία τμήματα. Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ως προς, την, ε, το δυναμικό, την ενδυνάμει δηλαδή πορεία μας και το δυναμικό που ενυπάρχει. Στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική κινητοποίηση. Σε ποιες τεχνολογίες βασίζεστε. Δεν διάβασα την έρευνα, όλη την έρευνα, αλλά ποια, ποιες προδιαγραφές προβάλλεται και στον τομέα των ε, ευρεσιτεχνιών. Υπάρχουν κοινέ ε, ευρεσιτεχνίες, υπάρχει υποστήριξη, υπάρχουν ταμεία, υπάρχουν πόροι. Πώς έχει αυτό το εγχείρημα της μεταφοράς τεχνολογίας. Μας είπατε ότι δεν ξέρετε ποια είναι η ποσοστιαία αναλογία της ε, μεταφοράς, μεταφοράς δηλαδή από τον ένα τομέα στον άλλον. Πώς ε, το έχετε ε, αντιμετωπίσει αυτό, μιλάτε για την έρευνα, για τη βιομηχανική συνεργασία. γιατί αυτή η ακαδημαϊκή παρουσίαση μας δίνει μια γενική εικόνα, αλλά όχι τον τρόπο λειτουργίας του όλου εγχειρήματος έτσι ώστε να ορίσουμε την ε, κατάσταση επιχειρησιακά, να δούμε πού υπάρχει έμπρακτα μία πρόπτικη και ποια αποτελέσματα μπορούμε να αναμένουμε από τον βιομηχανικό τομέα. Και τέλος, πώς θα πρέπει να ποσοστοποιήσουμε το όλο εγχείρημα είπε ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες στον εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό τομέα. Πώς κρίνεται όμως την ευρωπαϊκή θέση έναντι άλλων χωρών, όπως της είπα και την Κίνα, διότι η Volvo αγοράστηκε από μία κινέζικη ε, μάρκα που ασχολείται με είδη νοικοκυριού. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτές τις συνέργειες, πώς μπορούν ε, να προωθηθούν, ε, έχουμε κάποια καθυστέρηση σε αυτό το τομέα ή προτρέχουμε και ζητώ συγγνώμη για τη χιονοστιβάδα ερωτήσεων. Συνάδελφος ένα έχει να βάλει ερωτήσει και μετά θα απαντήσουμε σε όλα μαζί. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομο γιατί θα βασιστώ στις δύο περιβάσεις των συναδέλφων. Δεν θέλω να προσθέσω, αλλά να πω απλώ ότι βρισκόμαστε στα περιθώρια της οικονομίας. Δεν έχουμε περάσει το σωστό ορόσημο, γιατί αν δεν τοποθετήσουμε και τη σοδρομική βιομηχανία μαζί με την βιομηχανία και την αναφιολογική έχουμε ένα πρόβλημα. Θα πρέπει οι τρεις αυτές βιομηχανίες να ασχοληθούν στην ε, βασική έρευνα ιδίως στα σύνθετα ε, υλικά. Και ό,τι έγινε μέχρι στιγμής δεν ήταν σωστά ε, διατυπωμένο γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε έξω από την έρευνα που έγινε για κάποιο συγκεκριμένο τομέα για να έχουμε μια καλή εικόνα για το μακροπρόθεσμα. Και όταν ε, μιλάω για το περιθώριο της οικονομίας βλέπουμε ένα σημαντικό ε, φαινόμενο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι έρευνες θέλουμε γιατί εάν το κύριο σημείο παραμένει το κόστος της εργατικής χείρας μπορούμε, δεν θα προχωρήσουμε γιατί όλες οι μεγάλες βιομηχανίες πηγαίνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή τη στιγμή η Ρενό επενδύει στην Ρουσία εκατοντάδες εκατομμυρίων ε, ευρώ σε ένα τεράστιο βιομηχανικό κέντρο και μετά επανεισαγάγει τα οχήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την αεροναυτική το πρόβλημα είναι ακόμη πιο μεγάλο. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Μπορεί να κάνουμε ε, οικονομία στην έρευνα και σε τι χρησιμεύει αυτό όταν η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία ή οι κάτω χώρες χρηματοδοτούν το F-35 που οι ε, Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας δολοφόνος της, Ευρωπαϊκή της ευρωπαϊκής αερονομικής βιομηχανίας. Τι βοηθάει όταν οι ε, Κινέζοι χρηματοδοτούν έναν ανταγωνιστή του 320 παραδείγματο χάρη. Μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Χρειάζομαι όμως να περάσουμε από αυτά για να φροντίσουμε η δική μας παραγωγή να είναι αναγνωρισμένη και σεβαστή. Γιατί εμείς δεν έχουμε πάντα τους ίδιους περιορισμούς όσον αφορά την παραγωγή. Και το κύριο θέμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συζήτηση για την έκθεσή σας είναι ένα ουσιαστικό θέμα η γενιά της baby boom θα περάσει στην, ε, ε, στη σύνταξη προσεχώς. Τι θα γίνει να, για να αντικαταστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στήριζαν την αεροφυγική βιομηχανία στην Ευρώπη. Πρόεδρος, τώρα θα σας ήμουν ευγνώμων εάν απαντούσατε σε ερωτήσεις και εάν απαντούσατε πολύ σύντομα μάλιστα. Σε σχέση με τις βιομηχανίες που ανέφερε η κυρία Τροτμάν, σε αυτή τη μελέτη ενεπλάκησαν διαφορετικές εταιρείες. Παραγωγή εξαρτημάτων και δομικών λίθων των αεροσκαφών και των αυτοκινήτων. Επίσης και από τον πανεπιστημιακό τομέα είχαμε παρουσία, όπως είχαμε και παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από τους δύο τομείς. Και είχαμε ακριβώς όπως ελέγχθη την ανάδραση από τους διάφορους φορείς της Ενώσης που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και ορισμένα ερευνητικά συμπλέγματα που έχουν γνώμη για τους δύο αυτούς τομείς. για τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Η μελέτη μας είναι ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια εντοπισμού των συνεργειών. Η άποψη των περισσότερων εμπλεκομένων ε, φορέων ήταν ότι μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες <clears throat> δράσεις οι οποίες να ευνοούν την συνέργεια στις περιοχές που εντοπίσαμε εμείς ως υψηλής, υψηλού δυναμικού. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες εργάζονται και οι δύο <clears throat> τομείς. Και είναι φυσικά αρκετά δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσουν να συνδυαστούν, γιατί είναι διαφορετικές οι απαιτήσει στους δύο τομείς. Είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει η μεταφορά της τεχνολογίας. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ερευνών. Επομένως αυτή η έρευνα είναι αυτό το οποίο μπορούσε να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές της τελευταίας πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος του πρόγραμματος πλαισίου 7, αν υπήρχε παραγωγή χάρη μια πρόσκληση για την ε, ε, έρευνα στην χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε διαφόρους τομείς, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια εκκίνηση για να κάνουμε περαιτέρω έρευνες. Τι άλλες προσπάθειες θα πρέπει να προβλέψουμε για το μέλλον. Είναι το ερώτημά σα. Πιστεύω ότι αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο θέλουν οι τομείς αυτοί να προχωρήσουν περισσότερο. Οι ίδιοι αυτοί οι τομείς είναι αυτοί οι οποίοι, οι οποίοι θα πρέπει να εμπλέκονται πλήρως 100% σε αυτούς τους τομείς. Για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο πιστεύουμε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 για την έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να δώσει πολύ περισσότερο χώρο, πολύ περισσότερες προσπάθειες <clears throat> για να προωθήσει προγράμματα τα οποία θα είναι κοινά μεταξύ και των δύο τομέων, μάλλον να κάνει υποχρεωτικό να εμπλέκονται και οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι και από τους δύο φορείς, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορέσουν να εξασφαλιστούν κοινέ προδιαγραφές και για τους δύο τομείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν δεν έχω λησμονήσει κάτι, έχω απαντήσει. Και ίσως θα μπορούσα να κάνω και κάποια παρατήρηση για τα σχόλια της συναδέλφου μου. Είναι μια πρώτη μελέτη. Αυτό το οποίο θέλαμε να ξέρουμε είναι αν είχε νόημα ή όχι να προχωρήσουμε σε αυτή την αναζήτηση συνεργειών και αν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να υπάρξει μεταλαμπάδευση τεχνολογίας μεταξύ <clears throat> δύο διαφορετικών τομέων, αυτοκινήτου και αεροσκαφών. Για τις λεπτομέρειες που χάρη των υλικών, το αν είναι παραγωγός χάρη δομικά υλικά με ενίσχυση από νανοίνες, αν είναι πιο ε, ικανά να απορροφούν ενέργεια, θόρυβο και αν είναι πιο ισχυρά ή όχι. Όλα αυτά τα θέματα είναι καλύτερο να τα θέσετε στις πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την έρευνα για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν επιτροπές οι οποίες υπάρχουν ήδη μέσα στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος καθορισμός της θεματικής, πιο συγκεκριμένα από ό,τι κάναμε εμείς και εμείς φυσικά δεν είχαμε ακριβώς αυτό το στόχο να υποκαταστήσουμε αυτές τις επιτροπές. Πιστεύω ότι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν και αυτή είναι μία από τις συστάσεις μας να, είναι, να υπάρχει πραγματικά συγκεκριμένη διατύπωση τέτοιων είδων προσκλήσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δύο αυτά θέματα, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε και τους δύο να είναι παρόντες στο ίδιο τραπέζι και να γίνεται παντού αυτή η μεταλαμπάδευση, αλλά είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η συνέργεια. Για το πώς θα εφαρμοστούν αυτά σε βιομηχανικό τομέα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Για τον κύριο Ενέν, μιλήσατε για εξοικονόμηση σε ό,τι αφορά την έρευνα και ανάπτυξη. Εμείς δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό, προφανώς είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η εξοικονόμηση. Εμείς θέλουμε να έχουμε περισσότερη έρευνα και, και ανάπτυξη. Αυτό το οποίο εμείς αναζητούμε είναι η βελτιστοποίηση της έρευνας και της ανάπτυξης και όχι η εξοικονόμηση χρημάτων για τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πολλές ερωτήσεις υποβλήθησαν, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, που μας κάνετε την παρουσίαση. Ευχαριστώ και συναδέλφου. όσοι τουλάχιστον άνοιξαν μέχρι το μέλλον. <laughs> Τέλος, σας εύχομαι καλό βράδυ. Θα ξαναδεθούμε αύριο το πρωί και συνέχιση της μας. Καλό βράδυ.